Καλησπέρα σα. Ε, θα ήθελα πριν να προχωρήσουμε στην ε, ημερήσια διάταξη να ε, σας κάνω μια ανακοίνωση. Σύμφωνα με τους συντονιστές, με την απόφαση των συντονιστών, θα χρειαστεί να ψηφίσουμε σε σχέση με τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουμε όσον αφορά τις Αναφορές για το Πακιστάν. Ξέρετε ότι ενευλήθη πέρυσι λόγω της απαραίτητης εξαίρεσης που έπρεπε να δοθεί από τον ΠΟΕ. Θα πρέπει λοιπόν να ζητήσουμε από την Ολομέλεια μια εντολή ώστε να μπούμε σε άτυπο τρίλογο τριμερή διάλογο με το Συμβούλιο για αυτό το θέμα για να μπορέσουμε να έχουμε μια συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση. Εν τω μεταξύ, η Κομισιόν θα κάνει άτυπη σύσκεψη με το Συμβούλιο για να προετοιμάσει το τριμερή διάλογο. Αυτό αποφασίστηκε. Επίσης, αποφασίσαμε να διευρύνουμε την προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών σε σχέση με την έκθεση Hackard Να παρατείνουμε δηλαδή με δύο μέρες μετά από την αναμενόμενη λήψη απόφαση στην ΑΦΕΤ. Του ζητήσαμε λοιπόν να παραταθεί η δική μας προθεσμία. Η προθεσμία ήταν μέχρι που δεν θυμάμαι πότε. Could you tell me? What was the deadline? deadline on uh, Ποια ήταν η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών για την ΆΚΑ. Οκ, there Α, δεν υπήρχε πρόγραμμα. Ωραία, λοιπόν, τώρα όμως υπάρχει. Έχουμε δύο μέρες μετά την λήψη της απόφασης από την ΑΦΕΤ. Και θα σας ενημερώσουμε όταν θα γίνει αυτό. Ας προχωρήσουμε στο σημείο 8. Μάλλον, περαιτέρω ανακοινώσει. Το σημείο 18 θα αναβληθεί. Επρόκειτο για την παρουσίαση μια μελέτης για την πρόσβαση της προσχώρηση της Ρωσία στον ΠΟΕ και τι επιπτώσει αυτού για τις οικονομικές σχέσεις μεταξύ Ένωση και Ρωσία. Διότι ο συντάκτη αρρώστησε. Ε, Οπότε τώρα ας ε, συνεχίσουμε, συνεχίσουμε τις εργασίες μας. Για το σημείο 17 Το σημείο 14 αφορά τη συμφωνία ε, για το εμπόριο εξαρτημάτων και κατασκευαστικών στοιχείων μηχανοκίνητων οχημάτων. Το 15 η συμφωνία για τη διατήρηση των δεσμεύσεων για τις συναλλαγέ στον τομέα των υπηρεσιών. Ο εισηγητή είναι ο Τζαν Λούκα Σούστα. 16, το σημείο 16 είναι η συμφωνία με τη Ρωσία για την εισαγωγή, την αύξηση από τη Ρωσική Ομοσπονδία των Εξαγωγών Δασμών επί των πρώτων υλών. Η συγγήτρια είναι ε, και ο συγγητής είναι η Νέζε Βάιντερε. Και τέλος έχουμε τη συμφωνία πάλι με την Ρωσία για τη διαχείριση των δεσμολογικών ποσοστώσεων που εφαρμόζονται στις εξαγωγές ξυλίας. Η συγγητής Νέζε Βάιντερε. Η κυρία Νέζε Βάιντερε. Θα αρχίσω δίνοντας το λόγο στους εισηγητές, εάν είναι παρόντες. Ε, ισχύει για τον κύριο Ζαλέσκι που είναι ο πρώτο ε, και βρίσκεται εδώ στο έδρανο τη Προεδρία γιατί είναι αντιπρόεδρο τη Επιτροπή. Έχει το λόγο. Πάβελ. Ευχαριστώ πολύ Βιντάλ. Θα μιλήσω πολωνικά. Κάποιες παρατηρήσεις. Καταρχήν μιλάμε για μια συμφωνία που αφορά την προσχώρηση της Ρωσίας στον ΠΟΕ. Πράγμα το οποίο από μόνο του είναι πολύ θετικό και αναμένεται εδώ και πολύ καιρό από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ούτως, γιατί αυτή η προσχώρηση θα βελτιώσει και τις εμπορικές και οικονομικές σχέσεις μεταξύ Ρωσίας και ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, όμως ο προβληματισμός αφορά το κόστος που θα επιβαρύνει με το οποίο θα επιβαρυνθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θα πρέπει να πω ότι οι παραχωρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τη Ρωσία αφορούν για παράδειγμα τη συμφωνία για το εμπόριο εξαρτημάτων και στοιχείων μηχανοκίνητων οχημάτων. Πρόκειται για μια πραγματική άδεια παραχώρηση και είμαι ευτυχή και ευγνώμων προ την Κομισιόν, γιατί σήμερα μπορούμε ει βάθο να συζητήσουμε όλα αυτά τα ζητήματα. Και άρα θα μπορέσουμε να συζητήσουμε <clears throat> και για τις συνέπειες που θα προκύψουν τη στιγμή που η Ρωσία θα προσχωρήσει στον ΠΟΕ. Ακριβώς αυτό είναι το ευρύ πλαίσιο επί το οποίο θα πρέπει να ε, εκφέρουμε άποψη και να αποφασίσουμε αν θα δώσουμε τη σύμφωνη μας γνώμη. Για την ώρα η θέση της Κομισιόν προσπαθεί κάπως να καθησυχάσει όλους, καθώς λέει ότι οι συνέπειες για όλους τους εμπορικούς τομείς θα είναι θετικές και συμφέρουσες. Και λέει μάλιστα ότι έχει προβλεφθεί και έχει γίνει αντικείμενο διαπραγμάτευσης και ένας μηχανισμός ε, ε, ασφαλείας. Οπότε αν υπάρξει μια μεγάλη πτώση των ευρωπαϊκών εξαγωγών προς τη Ρωσία θα αρχίσει αυτόματα να ισχύει. Και με αυτόν τον τρόπο θα καταφέρουμε να αποφύγουμε μια υπερβολική αποδυνάμωση των ευρωπαϊκών εξαγωγών προς τη Ρωσία. Όλα αυτά έχουν πολύ μεγάλη σημασία γιατί ο αυτοκινητο, η αυτοκινητοβιομηχανία και ο κλάδος της είναι ένας από τους πιο σημαντικούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από την άλλη πλευρά, οι παραχωρήσεις ε, που έχουμε πετύχει από την, ε, μάλλον που δίνονται στη Ρωσία, ε, είναι πολύ σημαντικές. Κατά συνέπεια, θα ήθελα τελειώνοντας να πω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να παρακολουθεί διαρκώς ε, τις εμπορικές ανταλλαγές, ε, ούτως ώστε ε, τη στιγμή που θα υπάρξουν εμπόδια στην εφαρμογή του μηχανισμού ασφαλείας να ξεπεραστούν μέσω της άμεσης λειτουργίας του μηχανισμού ασφαλείας. Επίτα θεωρώ ότι η υιοθέτηση αυτού του πακέτου θα πρέπει να εξαρτηθεί ή να, να συνδεθεί από τα πλεονεκτήματα και τις συνθετικές συνέπειες που θα προέλθουν από την προσχώρηση της Ρωσίας στον ΠΟΕ και από τις παραχωρήσεις που θα δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι σημαντικό να έχουμε όλες τις ε, πληροφορίες που πρέπει ώστε να μπορούμε να αποφασίσουμε όριμα. Σας ευχαριστώ. Έχουμε λοιπόν και συζητάμε το, τις εμπορικές ε, σχέσεις της ίδιας. Σας περάσουμε στη δεύτερη έκθεση. Εδώ έχουμε συγητή τον κύριο Σούστα. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Όπως ε, ήδη θυμήσατε, αυτές οι συμφωνίες εντάσσονται στο πλαίσιο της προσχώρησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Παγκόσμια Οργάνωση Εμπορίου μετά από 18 χρόνια Απόπειρε. Είναι σημαντικό γεγονός για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά πάνω απ' όλα για τη Ρωσία. Αλλά πιστεύω πως πάνω απ' όλα σημαίνει σημαντικές προοπτικές για τη δικιά μας κοινότητα. Μια αγορά υπό επέκταση και ανάπτυξη. 25% των εξαγωγών μας είναι υπηρεσίε προς τη Ρωσία και αυτή η συμφωνία να βελτιώσει μόνο θα μπορούσε ένα πλαίσιο που ήδη είναι σημαντικό. Σε ορισμένου τομεί οι δεσμεύσει φαίνονται να είναι πιο σημαντικέ, όπω στον τομέα των τηλεπικοινωνιών ή των ε, χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, ενώ σε άλλου τομεί φαίνεται να είναι πιο χαμηλέ οι δεσμεύσει για δραστηριότητε ε, που αφορούν ξένες επιχειρήσεις. Η Ρωσία μέσω αυτής της συμφωνίας, μέσω αυτών των συμφωνιών αποφάσισε να καταρρύψει φραγμούς και να δώσει μια πιο ευνοϊκή αντιμετώπιση στους ξένους επενδυτές σε 11 τομείς που συμπεριλαμβάνουν 118 υποτομείς, υπηρεσίες, ε, οικοδομικές υπηρεσίες, ε, ταχυδρομικές υπηρεσίες, τηλεπικοινωνίες, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες κτλ. Είναι σημαντικό πλαίσιο και θα πρέπει στην πράξη να να επαληθεύσουμε αν όντω τηρούνται οι υποσχέσεις της Ρωσίας τόσο στο επίπεδο εφαρμογής των κανόνων που ισχύουν για τις ε, ανηλυμένες αυτές υποχρεώσεις όσο και σχέση με την ε, μεταρρύθμιση της ρωσικής νομοθεσίας για το άνοιγμα της αγοράς. Τώρα, όσον αφορά τη συγκεκριμένη συμφωνία για τη διατήρηση των δεσμεύσεων για τι συναλλαγέ στον τομέα των υπηρεσιών, περιέχονται στη σημερινή συμφωνία, ε, θα πρέπει να πούμε ότι έχουμε μια συμφωνία που σχετίζεται με τις ε, διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές και τις προσωρινές μετακινήσεις ε, προσωπικού για επαγγελματικούς λόγους και οι δεσμεύσεις της Ρωσίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι παραπάνω από αυτές που έχει να αναλάβει η Ρωσία στο πλαίσιο του ΠΟΕ. Άρα λοιπόν έτσι ώστε να διατηρηθούν οι συνθήκες αυτές έχει υπογραφεί μια διμερή συμφωνία που στόχο έχει να διατηρήσει τα πλεονεκτήματα και τα προνόμια της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς να υπάρχει αυτή η λογική της ε, Ανταλλαγή ή της επιστροφής απέναντι στη Ρωσία, απέναντι στην οποία δεν έχουμε αναλάβει νέε ε, ε, δεσμεύσεις. Γι' αυτό και είναι σημαντικό να επαναλάβουμε το γενικό θετικό αντίκτυπο και το θα, ε, για, όσον αφορά την σύνδεση της Ρωσία με τον ΠΟΕ και την βούληση της Ευρωπαϊκής Ένωση να ολοκληρώσει τη διμερή συμφωνία που περιλαμβάνει επιπλέον όρους σε σχέση με το γενικότερο πλαίσιο ε, στον τομέα των υπηρεσιών. Τώρα, σε σχέση με την νέα διμερή συμφωνία εταιρική σχέση με τη Ρωσία, θα πρέπει να υπογραμμίσουμε παλιές ε, υποχρεώσεις για να αποφύγουμε για να, μάλλον, να θυμίσουμε τα κεφάλαια 3 και 4 που αφορούν το εμπόριο και τις υπηρεσίες προς επιχειρήσεις. Είναι ένα κείμενο ε, με το οποίο συμφωνούμε και οι περαιτέρω βελτιώσεις που θα επιφέρουμε θα το καταστήσουν ακόμα καλύτερο. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστούμε Τζαν Λούκα τώρα για τις επόμενους δύο φακέλους. Είναι η, κυρία, η η κυρία ε, Ινέζε Βάιντερ από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Δεν θα επαναλάβω το περιεχόμενο και τη συλλογιστική που διέπει δύο εκθέσεις ε, για τη Ρωσία και για τι πρώτε ύλε, διότι τα έχουμε συζητήσει σε προηγούμενη συνάντηση. Αναγνωρίζουμε τη σημασία και το κατεπήγον των δύο φακέλων, γι' αυτό και πρότεινα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να δώσει σύμφωνη γνώμη. Ωστόσο, θα ήθελα να κάνω κάποιε παρατηρήσει για κάποιες ελλείψεις και μετά από τις ερωτήσεις που αποφθήναμε στην Κομισιόν. Πρώτα απ' όλα, η Συμφωνία για τις πρώτες ύλες, για να τα πω και τα δύο μαζί. Ξεκινάω πρώτα από τη Συμφωνία για τις πρώτες ύλες. Όπως γνωρίζετε, είναι συμπληρωματική προς τις δεσμεύσεις ε, της Ρωσίας ε, προς τον ε, ΠΟΕ. 700 προϊόντα, πρώτες ύλες, έλαια, πετρέλαιο κτλ. Όλα αυτά είναι περίπου το 80% των βουναπρώτων υλών που εξάγει η Ρωσία και για το οποίο θα υπάρχουν πλέον δεσμευτικοί δασμοί. Όπως έχω πει και στην ετολογική έκθεση της εκθέσή μου, αυτό που με ανησυχεί κυρίω εδώ είναι ότι δεν είναι πολύ συγκεκριμένη η διατύπωση το να καταβληθούν οι βέλτιστες προσπάθειες ε, και να υπάρξει διαβούλευση αυτό δεν αρκεί γιατί θα μπορούσε να συνεχίσει η Ρωσία να ε, χρησιμοποιεί τα προστατευτικά μέτρα που έχει χρησιμοποιήσει επί σειρά ετών. Θα πρέπει λοιπόν ε, να προσέξουμε τη διατύπωση για να είναι επιτυχημένη αυτή η συμφωνία και ιδίως να δούμε τι συμβαίνει σε περίπτωση που δεν τηρεί η Ρωσία μια από τις προτάσεις. Τι κάνουμε στη διάρκεια της διαδικασίας διαβούλης που προβλέπετε, τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν βλέπω και πολλά εργαλεία μέσω των οποίων θα μπορούσαμε εμείς να επιβάλλουμε την συμφωνία αυτή, ιδίω γιατί υπάρχουν κάποια πράγματα που δεν συμπεριλαμβάνονται στη συμφωνία σύνδεση, μάλλον ένταξης της χώρας στον ΠΟΕ. Πώ μπορούν να μπουν λοιπόν ε, οι ρήτρε για την εφαρμογή μηχανισμών επίλυσης διαφορών σε αυτέ τι περιπτώσει. για Τώρα έρχομαι στο δεύτερο θέμα που είναι η αύξηση των εξαγωγικών δασμών επί των πρώτων ε, υλών για τα προϊόντα. Ξυλίας. Μιλάμε για την ε, μάλλον για τις ποσοστώσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαχειρίζεται εδώ ποσοστώσεις εξαγωγών πρέπει να υπάρχει ένα ρυθμιστικό πλαίσιο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει κάποιες διτάξεις και συγκεκριμένα μια εφαρμοστική πράξη. Αλλά φαίνεται να υπερβαίνονται οι διατάξεις του ΑΡΤ 218 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήταν ίσως καλύτερο να γίνει μία πράξη συναπόφασης, 207 άρθρο δηλαδή, και να συμμετέχει και το Κοινοβούλιο. Τη Δευτέρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχολίασε ότι η υλοποίηση των εξαγωγικών ποσοστώσεων θα γίνεται σε βάση όποιο έρχεται πρώτος εξυπηρετείται πρώτος. Δεν απαιτείται δηλαδή ατομική μεμονωμένη απόφαση από την ε, εφαρμοστική αρχή και δεν θέλει να τροποποιήσει, να προσθέσει κάτι η Κομισιόν. Όμω τέτοιε νομοθετικέ διατάξει ε, βλέπουμε ότι προτείνονται ιδιαίτερα σε διάφορε συμφωνίε διεθνού εμπορίου. Φαίνεται να είναι όλο και αυξανόμενη αυτή η τάση. Ελπίζω λοιπόν στο μέλλον οι εν λόγω διατάξει δεν θα ε, περιλαμβάνονται πλέον σε προτάσεις για επερχόμενες ε, συμφωνίες και σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου. Ευχαριστώ. Thank you. So we have uh, the presentation. Ακούσαμε λοιπόν τις παρουσιάσεις από τους εισηγητές των τεσσάρων σχεδίων σύστασης. Πρέπει να δώσουμε σύμφωνη γνώμη για τις ε, συμφωνίες αυτές και ξεκινά τώρα η συζήτηση. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος που θέλει το λόγο. Μπεν Λάγκε. in Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Βρίσκω τις εκθέσεις, τις εκθέσεις σας πραγματικά καλές και αντανακλούν το γεγονός ότι κατ' ουσία ε, πρόκειται να συμφωνήσουμε με τις συμφωνίες αυτές, ε, να δώσουμε τη συγκατάθεσή μας. Βεβαίως υπάρχουν κάποια σημεία τα οποία δεν μπορούμε να αποδεχθούμε. Και για να επανέλθουμε στη συμφωνία για την αυτοκίνητη αυτοκινητοβιομηχανία, κατ' ουσία όταν προσχωρεί κανείς στο ΠΟΕ, αυτό σημαίνει ότι ισχύουν οι ίδιοι κανόνες. Και τώρα θέλουμε να δημιουργήσουμε στην περίπτωση αυτή ένα δίκτυο ασφαλείας, γιατί δεν ξέρουμε κατά πόσο η άλλη πλευρά πρόκειται να τηρήσει τους κανόνες του παιχνιδιού. Και πράγματι μπορούμε να θέσουμε το ερώτημα κατά πόσο το επενδυτικό πρόγραμμα στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας στη Ρωσία ανταποκρίνεται στις συνήθειές μας όσον αφορά το δίκαιο για τις επιχορηγήσεις. Και εδώ έχω κάποια προβλήματα και το ερώτημα είναι κατά πώς θα πρέπει να γίνει μια επέκταση μέχρι το 2018. Και αν θέλουμε να έρθουμε στην έκθεση για τις πρώτες ύλε, τότε θεωρώ ότι ακόμα και ο ίδιος ο τίτλος είναι κάπως ε, εντυπωσιακός. Δηλαδή, Εάν κινείται κανείς στο πλαίσιο του ΠΟΕ, θεωρεί κανείς ότι οι τελωνιακοί δασμοί καταργούνται, αλλά και δεν διατηρούνται και ούτε καν βεβαίως αυξάνονται. Άρα λοιπόν εδώ ενέχεται μία αντίφαση όσον αφορά την αξίωση κοινών, θέσπιση κοινών κανόνων στο πλαίσιο του ΠΟΕ και ισχύω κοινών κανόνων. Τώρα, Όσον αφορά τις προσπάθειες της ε, Ρωσίας για την μείωση, ενδεχομένως αυτός ο κατάλογος των 700 ε, τομέων είναι εξαντλητικός. Δηλαδή, δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι αν ε, ξαφνικά θεωρηθούν ενδιαφέρουσες κάποιες άλλες πρώτες ύλες θα συμπεριληφθούν και αυτές στον κατάλογο. Όχι, αυτό δεν επιτρέπεται να συμβεί σε καμία περίπτωση. Και άλλωστε σε αυτό αναφέρθηκε και η ίδια η συγγήτρια. Ε, πόσο ισχυρές είναι οι δεσμεύσεις. Δηλαδή όταν διαβάζουμε τη φράση κάνουν τις ε, ε μεγαλύτερες δυνατές προσπάθειες κλπ. Όλα αυτά δεν έχουν καμία δεσμευτικότητα και κατ' ουσία σχετικοποιούν τις διατάξεις. Τώρα όσον αφορά δηλαδή τις πρώτες ύλες, μπορούμε ε, γενικά να το αποδεχτούμε μόνο εφόσον ε, τεθεί ένας χρονικός περιορισμός. Και τελικά η αντιμετώπιση του ζητήματος των πρώτων υλών καταλήξει σε μια δεσμευτική συμφωνία με ενιαίους κανόνες. Ούτε ώστε να μπορεί κανείς να είναι βέβαιος ότι μελλοντικά αποκλείεται να ένα το κόστος για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και στην τελευταία έκθεση που αφορά την ξυλία, και εδώ μπορεί κανείς να θέσει το εξή ερώτημα. Χρειαζόμαστε μια ρύθμιση επί τη βάση ποσοστώσεων ή δεν θα έπρεπε στον ΠΟΕ να υπάρχει μια απελευθέρωση του εμπορίου. Και αν θέσει κανείς επιτάπητο στο ζήτημα των ποσοστώσεων, βεβαίω τότε ακολουθεί το ερώτημα ποιος έχει κατ' ουσία το δικαίωμα να αποφασίζει για τις ποσοστώσεις. Θέμα το οποίο αφοράπτεται του δικαιώματος απόφασης του Κοινοβουλίου, το οποίο τίθεται να αμφιβόλο. Και με τον τρόπο αυτό περιορίζονται οι στην απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Άρα θα έθετα εδώ το εξής ερώτημα τέτοιου είδους ε, ρυθμίσεις δεν είναι δυνατόν να έχουν μια ηγετική θέση στο μέλλον. Ε, γιατί τελικά αφήνουν ανοιχτή την πίσω πόρτα για μια παράκαμψη των κανόνων. Παρ' όλα αυτά δεν θα αρνηθούμε την συγκατάθεσή μας. Είμαι σίγουρη ότι η Επιτροπή θα θέλει να πάρει θέση. Υπάρχει κανείς άλλος ομιλητής σε σχέση με το πακέτο για τη Ρωσία. Όχι. Τότε θα περάσουμε στην Επιτροπή. Έχουμε εδώ τον Πίτερ ε, Πάλας. Σας ευχαριστούμε πολύ και σας παρακαλούμε να σχολιάσετε τα όσα ακούσατε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, χαίρομαι πολύ που επέστρεψα σε μια τόσο σημαντική ευκαιρία που ελπίζω θα έχουμε μια θετική έκβαση για αυτές τις διμερείς συμφωνίες. Καταρχήν θα ήθελα να κάνω κάποια σχόλια γενική φύσεως. Καταρχήν σε σχέση με το ζήτημα που έθεσε ο κ. Ζαλεύσκη δηλαδή ότι συνολικά για όλα τα μέλη του ΠΟΕ είναι ευεργετικό να είναι ευεργετική η προσχώρηση της Ρωσίας στον ΠΟΕ και για την Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι υπαριθμόν ένα, ένα εμπορικός εταίρος της Ρωσίας, κάτι τέτοιο είναι ιδιαίτερος ευεργετικό. Ας μην ξεχνάμε που βρισκόμαστε σήμερα. Σήμερα έχουμε μία μάλλον αδύναμη διμερή συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ρωσίας που ανέφερε άλλωστε και ο κύριος Σούστερ η οποία ωστόσο δεν διατυπώνει ξεκάθαρες δεσμεύσεις εκ μέρους της Ρωσίας. Είναι μια άνηση συμφωνία. Εμείς ε, είμαστε δεσμευμένοι λόγω των δεσμεύσεων που έχουμε αναλάβει στο πλαίσιο του ΠΟΕ έναντι της Ρωσίας να της παράσχουμε την πιο, ευνοούμενη, την πιο ευνοϊκή ε, ε, μεταχείριση ενώ η Ρωσία δεσμεύεται τελικά να μας δώσει μόνο αυτό το οποίο δίνει και στους υπολείπους. Άρα λοιπόν η Ρωσία μπόρεσε το 2008-2009 να άρει ε, ευνηδίως τους ε, δασμούς για κάποια προϊόντα. Ήταν μέτρα για την αντιμετώπιση της ε, κρίσης και μπόρεσε να αυξήσει τις εξαγωγές της στη ξυλία και με τον τρόπο αυτό κατέστρεψε να κομμάτι της βιομηχανίας μεταποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σήμερα η Ρωσία μπορεί να χρησιμοποιεί τέτοια μέτρα ε, μη επιβολής ε, τελωνιακών ε, δασμών όσον αφορά για παράδειγμα την εισαγωγή αγροτικών προϊόντων. πέρσι ήταν το έτος των απορροκυπευτικών, φέτος είναι το έτος του κρέατος. Άρα λοιπόν οι Ρώσοι έχουν μια πραγματικά τεράστια φαντασία στην εξέβρεση λύσεων για, να, για την έξοδο από την κρίση. Και ε, ε, όσον αφορά την ε, διπλή επιβολή φόρων, κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατό και εάν η Ρωσία δεν τηρήσει τις δεσμεύσεις της μπορούμε να ε, την, ε, την αναγκάσουμε ε, μπορούμε να προσέξουμε μάλλον στο μηχανισμό επίλυσης διαφορών. Άρα λοιπόν δεν έχουν πλέον τις δυνατότητες που είχαν υπό την διμερή συμφωνία. Η Ρωσία κατά την άποψή μας έχει ένα υψηλής ποιότητας πακέτο προσχώρησης στον ΠΟΕ ε, σε, σχέση, σε σύγκριση με άλλες χώρες που έχουν πρόσφατα προσχωρήσει στον ΠΟΕ και ε, η σύγκριση αφορά μεγάλες οικονομίες όπως είναι η Σαουδική Αραβία, η Ουκρανία και κάποιες άλλες που προσχώρησαν στον ΠΟΕ τα τελευταία δέκα χρόνια και ασφαλώς είναι υψηλή ποιότητα σε σύγκριση με, τα προηγού, με τις προηγούμενες χώρες αναδυόμενες οικονομίες όπως είναι η Ινδία και η Βραζιλία που δεν έχουν ε, καμία δέσμευση σε σύγκριση με τη Ρωσία στην περίπτωση της Ινδίας ε, μπορούν να επιβάλλουν απαγορευτικούς ε, δασμούς σε μια σειρά ε, προϊόντων. Γιατί τα ιδρυτικά μέλη του ΠΟΕ την εποχή εκείνη δεν μπόρεσαν να επιβάλλουν κάποιους περιορισμούς. Για τη Ρωσία υπάρξει μια σημαντική αλλογή, γι' αυτό οι δασμοί θα, πέσουν, θα μειωθούν κατά 7 ή 8% ενώ της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιστοίχως είναι 4%. Δηλαδή ασφαλώς είναι υψηλότερη από ό,τι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και σε πολλούς άλλους τομείς όπως είναι οι υπηρεσίες και εκεί η Ρωσία έχει αναλάβει κάποιες δεσμεύσεις πολύ περισσότερο από άλλες αναδυόμενες οικονομίες και ε, όσον αφορά τις ε, προμήθειες, την προστασία ε, πνευματικής ιδιοκτησίας κλπ. Είμαστε πεπισμένοι ότι πρόκειται για ένα πακέτο το οποίο είναι επιτεύξιμο, αν θέλετε, στην παρούσα περίοδο. Τώρα, πέρα από τις ε, γενικές δεσμεύσεις, η Ευρωπαϊκή Ένωση διαπραγματεύτηκε πέντε επιμέρους συμφωνίες με τη Ρωσία που συζητώνται σήμερα. Τέσσερις από αυτές είναι νομικά δεσμευτικές. Η πέμπτη για τις πρώτες ύλες, ε, αποτέχουμε δεν είναι νομικά δεσμευτική έχει έναν πολιτικό χαρακτήρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υπέγραψε με τη Ρωσία πριν από 8 χρόνια, δηλαδή το 2004, τη διμερή συμφωνία που καλύπτει τους εξαγωγικούς ε, δασμούς για 700 προϊόντα, τα οποία είναι παλαιά προϊόντα, τα οποία την εποχή, στα οποία την εποχή εκείνη η Ρωσία επέβαλε εξαγωγικού δασμού. Για το καθένα από αυτά υπάρχει μια δέσμευση μείωση στι περισσότερε περιπτώσει, αλλά όχι πάντοτε που κατατείνει το 0 σε 4 έτη. Για άλλε πρώτε ύλε, η Ρωσία ήδη το 2004 δεν ήταν διατεθειμένη να αναλάβει καμία δέσμευση και είπε ότι δεν πρόκειται να επιβάλλει, δεν επιβάλλει εξαγωγικούς ε, δασμούς, αλλά θέλει να επιφυλάξει για τον εαυτό της τη δυνατότητα να επιβάλλει μελλοντικά κάποιους ε, δασμούς εφόσον συντρέχει λόγος, υποχρόν λόγος. Και με το σκεπτικό αυτό εμείς προσπαθήσαμε να αντλήσουμε το καλύτερο δυνατό από αυτές τις ε, πέντε συμφωνίες που είναι οι καλύτερες δυνατές συμφωνίες. Γιατί, όπως σας είπα, δεν υπήρξε εναλλακτική λύση. Εάν η Ρωσία ήταν διατεθειμένη πριν από 8 χρόνια να καταργήσει τους ελληνικούς δασμούς, τότε τα πράγματα ήταν διαφορετικά, γιατί θα ήταν δεσμευτικές οι συμμονίες αλλά υπάρχουν ε, και άλλες χώρες όπως η Ουκρανία που ανέλαβαν κάποιες ε, δεσμεύσεις για τους ε, τελωνιακούς δασμούς αλλά δεν τις στήρισαν πλήρως και νομίζω ότι ο κ. Λάγκεν ανέφερε ότι βεβαίως αυτό επιτρέπει μία απομάκρυνση από τους γενικά εφαρμοσιμούς εφαρμοστέους κανόνες του πω Και θα ήθελα να πω ότι δεν υπάρχουν τέτοιοι γενικά εφαρμοστέοι κανόνες. Γιατί όλες οι χώρες που προσχώρησαν τα τελευταία χρόνια, συμπεριλαμβάνονες και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν ένα περιθώριο ελευθερίας. Ακόμη και η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να θεσπίσει ε, εξαγωγικούς ε, δασμούς όπως η Ινδία, η Βραζιλία και πολλές άλλες. Η Ρουσία, η Ρωσία και η Ουκρανία, οι οποίες προσχώρησαν ακόμα πιο πρόσφατα, βρίσκονται σε ακόμα πιο πλεονεκτική θέση. Δεν θεωρούμε ότι πρόκειται για μια διακριτική μεταχείριση, αλλά είναι μια λογική αντίδραση εκ μέρους της Ευρωπαϊκής όσον αφορά την ε, εισαγωγή επιβολής ε, τελωνιακών ε, δασμών. Αυτό το οποίο ε, παίρνουμε ως αντάλλαγμα από τη Ρωσία ως πολιτική δέσμευση είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο δεν ισχύει για τους περισσότερους από τους άλλους εταίρους μας στον ΠΟΕ και βεβαίως μπορούμε να δούμε τις αρνητικές επιπτώσεις. Πολύ συχνά οι δασμοί αυτοί αυξάνονται και χωρίς να υπάρχει δυνατότητα νομικής ε, προσφυγής ε, εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί εμείς είμαστε μια εξαρτημένη εικόνα, ε, οικονομία, συγγνώμη, αγοράζουμε πρώτες ύλες και τις μεταποιούμε. Άρα λοιπόν πρόκειται για μια νομικά ισχυρή συμφωνία. Δεν ήταν δυνατόν να επιτευχθεί κάτι άλλο, γιατί η Ρωσία είπε ότι δεν είναι διατεθειμένη να εφαρμόσει κάποιες δεσμεύσεις. Αυτό που αποδέχτηκε είναι μία ρήτρα διαβούλευσης που μας παρέχει τα διπλωματικά μέσα για να χειριστούμε τέτοιου είδους καταστάσεις. Ε, και θα ήθελα να προσθέσω ότι η Ρωσία μέχρι τώρα δεν χρησιμοποίησε αυτή τη δυνατότητα, δηλαδή δεν αύξησε τους δασμούς ε, πέρα από την περίπτωση των 700 προϊόντων και στην περίπτωση που αυξήθηκαν οι δασμοί για την ξυλία υπό τους όρους της ε, προσχώρησης ε, δεν θα επιτρέψουμε στο 2007 αλλά σε ακόμα χαμηλότερα επίπεδα. Όσον αφορά τις θαλάσσιες υπηρεσίες και τις σχετικές συμφωνίες, δεν έχω να προσθέσω τίποτα στην πολύ καλή έκθεση του κ. Σούστερ. Θεωρώ ότι περιγράψατε πολύ καλά την κατάσταση την οποία επιθυμούμε να διατηρήσουμε ένα προτιμησιακό καθεστώς για την Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τις υπηρεσίες στον τομέα υπηρεσιών στη Ρωσία και αυτή είναι μια λύση παραπλήσια με αυτήν που υιοθετήσαμε για την Ουκρανία που έχουμε μια παραπλήσια διμερή συμφωνία. Και αυτό με οδηγεί στις τρεις υπόλοιπες συμφωνίες, ξεκινώντας με την έκθεση του κυρίου Ζαλεύσκη για την αυτοκινητοβιομηχανία. Και υπόθηκε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έδωσε κάποιες ε, παραχωρήσεις, έκανε κάποιες παραχωρήσεις στη Ρωσία, ε, υπογράφησε τη συμφωνία. Εγώ βλέπω τα πράγματα ακόμα διαφορετικά, γιατί η προσχώρηση στον ΠΟΕ είναι μονομερής διαπραγμάτευση. Τα μέλη του ΠΟΕ δεν ε, κάνουν παραχωρήσεις. Η προσχωρούσα χώρα αυτή η οποία αναλαμβάνει κάποιες δεσμεύσεις σε αντάλλαγμα για την προσχώρηση στο καθεστώς του ΠΟΕ και σε όλα τα ευεργεμετήματα από τα οποία εποφελείται. Στην περίπτωση της αυτοκινητοβιομηχανίας ε, αυτό το οποίο ισχύει είναι ότι η Ρωσία έχει μια μακρά επενδυτική, ε, έχει μια επενδυτική ε, πολιτική εδώ και πολλά χρόνια και εφαρμόζουν την πολιτική αυτή σε πολλούς τομείς, στη γεωργία, στις, στην κατασκευαστική βιομηχανία, στα φαρμακευτικά προϊόντα κλπ. Αυτό το οποίο διαπραγματευθήκαμε είναι ότι από τη στιγμή που προσχώρησαν στο ΠΟΕ, κάθε ένας ε, κάθε ένα από αυτά τα μη συνεκτικά μεταξύ τους ε, μέτρα που αφορούν τις επενδύσεις θα απαγορευτούν, γιατί μέχρι στιγμή μπορούσαν να τα εφαρμόσουν. Μπορούν να εφαρμοστούν μόνο στην περίπτωση της αυτοκινητοβιομηχανίας και αυτή είναι μια λύση η οποία γίνεται αποδεκτή από όλα τα μέλη από όλα τα άλλα μέλη του ΠΟΕ. Μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση ήθελε να διαπραγματευτεί μια επιπρόσθετη διμερή δέσμευση, δηλαδή εάν κατά τη διάρκεια αυτή τη περίοδου μέχρι το 2018 θα υπήρχε μια αρνητική επίπτωση στις εξαγωγές, στις εξαγωγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ανταλλακτικά και τα κατασκευαστικά ε, τμήματα τότε θα μπορούσε να ανασταλεί αυτή η συμφωνία. Αλλά θεωρώ ότι δεν θα χρησιμοποιηθεί αυτή, κατά πάσα πιθανότητα αυτή η ρήτρα διαφύλαξη, αλλά μπορεί να ενεργοποιηθεί εάν διαπιστωθούν αρνητικέ επιπτώσει για τι εξαγωγέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Από 25% λοιπόν θα περάσουμε, από 50% θα περάσουμε στο 25% και αυτό σημαίνει ότι τα, οι εξαγωγές αυτοκινήτων από την Ευρώπη προς τη Ρωσία που δεν παράγονται στη Ρωσία θα μπορούσαν να χαίρουν από αυτές τις, ε, αυτών των δεσμεύσεων. Τέλος, ε, τα περισσότερα, οι περισσότερες μεγάλες ευρωπαϊκές και αμερικανικές εταιρείες ήδη εδώ και χρόνια κάνουν επενδύσεις στη Ρωσία. Ε, ωφελούνται από τους κανόνες αυτούς, διότι έτσι δημιουργείται πιο ισότιμο πεδίο για τους επενδυτές σε σύγκριση με τους Ρώσους ε, κατασκευαστές αυτοκινήτων. Ε, για να είμαστε ειλικρινεί, λοιπόν έπρεπε η Κομισιόν να βρει μια ισορροπία ανάμεσα στα συμφέροντα των εγκατεστημένων επενδυτών και τα συμφέροντα των Ευρωπαίων εξαγωγέων. Για την ξυλία τέλος. Εδώ οι κανόνες του ΠΟΕ για τη Ρωσία, το καθεστώς του ΠΟΕ για τη Ρωσία είναι το εξής. Βασικά ισχύει εκτός ποσόστοσης, την οποία έχει διαπραγματευτεί πολύ ψηλά για τα, τους εξαγωγών, αυτό για τα κονοφέρα που είναι, κονοφόρα που είναι το μεγαλύτερο κομμάτι των ευρωπαϊκών συμφερόντων για τις εισαγωγές. Και εδώ έχουμε, το, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το μόνο μέλος του ΠΟΕ που έχει δική του, δική του ποσόστοση. Οι υπόλοιποι, τα υπόλοιπα μέλη του ΠΟΕ θα μπορούν να εισάγουν ξυλία σύμφωνα με τη γενική ποσόστοση. Αυτό που κάνει αυτή η συμφωνία είναι, λοιπόν εκτός που εξασφαλίζει δική ποσόστοση για την Ένωση, εξασφαλίζει επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα καθοδηγεί το καθεστώς των εξαγωγικών δασμών της, για τη Ρωσία, γιατί οι εξαγωγικοί δασμοί ορίζονται, εκδίδονται από τη Ρωσία, αλλά θα πρέπει να ακολουθούν την απόφαση των ευρωπαϊκών αρχών όσον αφορά την κατανομή των ποσοστώσεων. Χώρες που έχουν ατυχείς εμπειρίες με ορισμένα ρωσικά μέτρα, και νομίζω ότι η Λετωνία συμπεριλάβανε τις αυτές, γνωρίζουν πως η κατανομή των ποσοστώσεων μπορεί να έχει καταστεί μυστηριώδης. Με αυτή τη συμφωνία αυτά θα τελειώσουν και νομίζω ότι αυτή είναι και η μεγαλύτερη χρησιμότητα της συμφωνίας. Ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω να απάντησα στις, στα σχόλια σας. Μάλιστα. Μετά από αυτή την εκτεταμένη επανέλθουμε για τις ε, τελικές παρατηρήσεις των εισηγητών. Να ξεκινήσουμε και πάλι με τον Παύλ Ζαλεύσκη. Uh, uh, σας ευχαριστώ πολύ για τις επεξηγήσεις που μας δώσατε. Πράγματι, ξεκινήσαμε τις σχέσεις μας με τη Ρωσία από πάρα πολύ χαμηλό επίπεδο και επομένως ε, η ένταξη της ε, Ρωσίας ε, στον ΠΟΕ τους εκπολίτησε θα έλεγα πιο πολύ και έτσι έχουμε πιο ισορροπημένες πλέον σχέσεις. Εγώ μπορώ να δεχθώ αυτό που είπατε, ότι ίσως πρέπει διμερώς να θεωρήσουμε ότι αυτή η συμφωνία είναι καλή και αμοιβαίως επωφελής. Σε αυτό το πνεύμα ζητώ να στηρίξουμε τη λύση αυτή για την αυτοκινητοβιομηχανία. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ πιστεύω πως δεν υπάρχουν πολλά να προσθέσει κανείς. έγιναν οι παρατηρήσεις που ήταν να γίνουν και είναι σύμφωνες και με τα όσα είπε και ο κύριο Διευθυντή. Ευχαριστώ. Ινέζε Βάιντερ. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί έδωσε μια πλήρη εξήγηση. Βέβαια, στη διάρκεια της παρέμβασής σας ε, μπορώ να σας πω ότι ονειρεύτηκα κάτι. γιατί δεν θέλω να ακούω συνέχεια όλα αυτά τα ωραία για την ανεφόρον αγάπη με τη Ρωσία. Γιατί έτσι το ήθελε η Ρωσία, γιατί αυτούς τους όρους έβαλε η Ρωσία. Εντάξει, η Κομισιόν είναι η Κομισιόν, εμείς όμως είμαστε πολιτικοί και γι' αυτό λοιπόν έχω ένα όνειρο κι εγώ. Ονειρεύομαι να είναι, αυτή η Ευρωπαϊκή, να είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή που θα θέτει τους όρους και όχι η Ρωσία και να είμαστε περήφανοι για τους όρους που θέτουμε. Αυτό ήθελα να προσθέσω μόνο και ελπίζω πραγματικά ναι, στρατηγική εταιρική σχέση. Όταν έφτασα εγώ στο Κοινοβούλιο πριν από 8 χρόνια, ρώτησα γιατί η Ρωσία είναι στρατηγικό εταίρο και η Ουκρανία, για παράδειγμα, δεν είναι. Πήρα μια απάντηση από του αρμοδίου, η οποία μου έλεγε ότι έτσι το ήθελε η Ρωσία. Γιατί το ήθελε η Ρωσία. Ελπίζω αυτή η νέα συμφωνία, η στρατηγική εταιρική σχέση να είναι ένα έγγραφο που και εμείς θα μπορούμε πραγματικά να θέτουμε τους κανόνες μας. Αυτό ήταν το όνειρο που ονειρεύτηκα. Κατά τα άλλα, σας ευχαριστώ πολύ για τις εξηγήσεις που μας δώσατε. Well, Commission was again asked uh, <laughs> a Αφού ετέθησαν ερωτήματα στην Κομισιόν, πρέπει να δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο να απαντήσει. Όχι, δεν νομίζω, λέει κύριε Βαϊτή. Εγώ κυρία μου θα σας παρακαλέσω να δείτε ε, τα σχόλια στο ρωσικό τύπο για να δείτε τα περί, περιόριστης ανεφόρων αγάπης και ένταξης στον ΠΟΕ. Υπάρχουν, ξέρετε, πάρα πολύ σημαντικά παράπονα από τους Ρώσους και η ρωσική κυβέρνηση προσπαθεί να εξασφαλίσει και τους ε, διαβεβαιώνει ότι θα τους προστατεύσει από τις εκτός που θα έχει η απελευθέρωση μετά την ένταξη στον ΠΟΕ. Σε ό,τι αφορά τη στρατηγική εταιρική σχέση, δεν έχουμε στρατηγική εταιρική σχέση πλέον. Έχουμε ολοκληρώσει μια πλήρη συμφωνία ελεύθερου πορείου με την Ουκρανία. Αλλά με τις παρούσες συνθήκες δεν μπορεί να ε, ολοκληρωθεί, δυστυχώς. Αλλιώς οι σχέσεις μας θα ήταν πολύ πιο προχωρημένες με την Ουκρανία από ότι με τη Ρωσία. Νομίζω ότι αυτές οι χώρες από πολιτικής πλευράς ε, αποτελούν μια πρόκληση και από οικονομικής πλευράς βέβαια. Τώρα ποιος έχει να αγάπη, έρωτα προς τη Ρωσία ε, δεν ξέρω. Πάντως για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιφυλάσσομαι. Λοιπόν, χρονοδιάγραμμα. Κατάθεση τροπολογιών, αν έχετε να καταθέσετε καμιά τροπολογία. Δεν ξέρω αν κανένα ε, θα μπορούσε να καταθέσει το για να πει όχι σε αυτή την συμφωνία, να μην δώσουμε έγκριση δηλαδή. Αλλά τέλο πάντων, ε, δεν σα λέω καν τι προθεσμίε. Το Μάιο θα εγκρίνουμε στην Επιτροπή μα ε, και στην Ολομέλεια του Στρασβούργου τον Ιούλιο θα γίνει η συζήτηση και η ψήφιση πριν τι καλοκαιρινέ διακοπέ. Και τώρα κάνουμε ένα άλμα. Και έχουμε μια κοινή συζήτηση για μια ακόμη φορά πάνω σε τρία θέματα. Δημόσιες συμβάσεις είναι το βασικό θέμα. Γνωμοδοτήσεις είναι και οι τρεις Αρμόδια επιτροπή είναι Επιτροπή ΜΚΟ. Πρόκειται ανταλλαγή απόψεων για τις τρεις αυτές γνωμοδοτήσεις. Εισηγητής και για τις τρεις. Για το πακέτο των δημοσίων συμβάσεων, ο Τζανλούκα Σούστα και του δίνω μέσα στο λόγο. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αν και πρέπει να συντάξουμε γνωμοδότηση επί, των, επί της ουσίας εκθέσεως ναι, της ΣΥΜΚΟ, σίγουρα πρόκειται για ένα στρατηγική σημασία θέμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται για γνωμοδοτήσεις για τις δύο οδηγίες που, που τροποποιούνται για τους κατοικές προμήθειες και για τις τοπικές δημόσιες υπηρεσίες και τις σχετικές προμήθειες όσον αφορά την εκχώρηση αδειών. Δεν χρειάζεται να πούμε πόσο πολύ συνδέεται και αυτό το θέμα με εκείνο που είναι αντικείμενο της πρωτοβουλίας των Επιτρόπων Μπαρνιέ και Ντεγκούχτ για το άνοιγμα των εξωτερικών αγορών στις Ένωσης στα θέματα των κρατικών προμηθειών και πόσο είναι σημαντικό για το ευρωπαϊκό βιομηχανικό σύστημα να μπορεί να έχει πρόσβαση σε ανοιχτές αγορές και έτσι να αναγνωριστεί και μια αμοιβαιότητα η οποία σήμερα δεν αναγνωρίζεται πλήρως και μάλιστα σε ορισμένες περιπτώσεις όχι απλά δεν αναγνωρίζεται αλλά ε, στην ουσία ακυρώνεται σε σύγκριση με τα όσα εμείς κάνουμε για τις άλλες χώρες για το ίδιο θέμα των δημοσίων, ε, των κρατικών προμηθειών και των ε, ε, τοπικών δημοσίων υπηρεσιών. Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό τομέα που είναι από τους λιγότερο απελευθερωμένους και τους λιγότερο ρυθμισμένους πρέπει να κινηθούμε μέσα στο νέο πλαίσιο που είναι υποκαθορισμό, καθορίστηκε και το Δεκέμβριο και θα δούμε τις λεπτομέρειές του στο πλαίσιο του Διεθνούς Οργανισμού Εμπαρίου. Είναι δεσμευτικοί αυτή οι νέοι ε, κανόνες μόνο για 42 χώρες και μάλιστα σε ορισμένε περιπτώσεις πρόκειται για στρατηγικού εταίρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι έχουν πολύ περίπλοκους ε, κανόνες ε, σε σύγκριση με εμάς που είμαστε πιο ανοιχτοί. Ακόμα και εκείνοι οι οποίοι είναι πιο ε, σύμφωνοι μαζί μας συνήθως έχουν νομοθεσία πολύ πιο δύσκολη, περίπλοκη, με μεγάλα προβλήματα πρέπει να επιληθούν. Υπάρχουν λοιπόν έλλειψη ισορροπίας μεταξύ των χωρών της Ένωσης και των εξοκοινωτικών χωρών Πρέπει ωστόσο να αποφύγουμε να υποκύψουμε σε έναν πειρασμό προστατευτισμού, αμοιβαιότητα, προσοχή στους κανόνες. Δεν σημαίνει να πέσουμε στον παγίδα του προστατευτισμού. Έχουμε παρακολουθήσει τους τελευταίους μήνες, τελευταίες εβδομάδες εκτός ε, Ευρώπης με την ρήτρα που εισήχθη από τον Ομπάμα για το Buy American Act και για τις ε, θέσεις ε, που ακούστηκαν μέσα στην Ευρώπη κατά τη διάρκεια της γαλλικής προεκλογικής εκστρατείας όσον αφορά το προστατευτισμό. Ε, σίγουρα δεν είναι αυτός ο δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουμε, αλλά ναι, ασφάλεια και προστασία των κοινωτικών συμφερόντων, ναι. Πρέπει να δούμε λοιπόν ποια είναι τα σημαντικότερα θέματα, τα ορόσημα. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι οι κρατικές προμήθειες και οι τοπικές δημόσιες υπηρεσίες θα πρέπει να υπόκειται σε κριτήρια ελευθερίας πρόσβασης, ελευθερίας οικονομικής προτεραιότητας, αλλά θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη και πολύ σημαντικές κοινωνικές ρήτρε. πρέπει να δούμε ε, τα κριτήρια επιλογής των, συμβαλ, συμβασι, συμβαλωμένων ε, ε, ε, ευρύτερα δηλαδή κριτήρια και όχι μόνο η χαμηλότερη τιμή, αξίες κατοφλίου αλλά και πολύ μεγάλη προσοχή όσον αφορά τις πιο πλεονεκτικές προσφορές. Πρέπει να δούμε και τις πιθανότητες υπεργολαβίας που πολύ συχνά είναι υπό τον έλεγχο της εγκληματικότητα και να φροντίσουμε ώστε να δημιουργήσουμε ένα σύστημα ελέγχου για τις δραστηριότητες όλων των φορέων που εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης έρχονται στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να συμμετέχουν στον διαγωνισμό αλλά και για να στηρίξουμε το δικό μας οικονομικό σύστημα ε, ε, ώστε να επεκταθεί και στις άλλες αγορές. Θα πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη την ανάγκη ε, εκμετάλλευσης αυτής της τεράστιας ευκαιρίας ώστε να, μην υπάρχει, ώστε να υπάρχει ισορροπία στις, ε, στα κριτήρια, στις αρχές της ελευθερίας και της ισότητας που είναι βασικά στοιχεία για τη δική μας νομική νοοτροπία και πολιτισμό και ταυτόχρονα να αναθεωρηθούν οι ευρωπαϊκές οδηγίες και να εισηχθεί ένα, μια νέα οδηγία όσον αφορά την εκχώρηση αδειών ε, και όλα αυτά να μην ακυρώσουν τόσο όσο κάνουμε για να στηρίξουμε τον εξωτερική ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Δεν χρειάζεται να υπογραμμίσουμε την σημασία αυτού του νομοθετικού πακέτου για το οποίο προετοιμάζουμε τις ε, γνωμοδοτήσεις μας στην αρμόδια επιτροπή επί της ουσίας, δηλαδή την ΙΜΚΟ. Γιάρος Λαβαλέσσα, ζήτησε πρώτο το λόγο από το ΕΛΚΑ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι. Η Σκιώδη, η συγκήτρια, κυρία Χάσλικ, δεν μπορούσε να έρθει σε αυτήν την ε, σημερινή συνεδρίαση γιατί παρήσατε στην συνεδρία της Επιτροπής ΙΜΚΟ που γίνεται παράλληλα. Ήθελα όμως να σας μεταφέρω κάποιες από τις παρατηρήσεις της. Η εξασφάλιση του κατάλληλου νομικού πλαισίου θα είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να υπάρχει διαφάνεια και για να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον φιλικό προς ε, συμπράξει δημόσιου ιδιωτικού τομέα, ιδίω σε διαφορέ σημαντικέ υποδομές. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για τις σχέσεις που εμείς έχουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση με τρίτες χώρες ε, όταν υπάρχουν εμπορικοί φραγμοί και μη ευνοϊκές ε, προϋποθέσεις και όροι νομικοί που επηρεάζουν αρνητικά. Επηρεάζουν και το εμπόριο και τις υπηρεσίες και τις δημοσίες συμβάσεις. Ε, οι συμβάσεις και η εσωτερική αγορά αλληλοσυνδέονται μεταξύ τους. Οι νομοθέτες, οι όσοι διαπραγματεύονται στο πλαίσιο του διεθνού εμπορίου θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τι διμερεί επιπτώσει που θα μπορούσαν να υπάρξουν και για την εσωτερική αγορά και για το διεθνέ εμπόριο. Και θα πρέπει να ακολουθήσουν μια συνεκτική προσέγγιση ώστε ο στόχος να είναι η προώθηση των ευρωπαϊκών αξιών, δηλαδή διαφάνεια, καταπολέμηση της ε, διαφθοράς, στήριξη των κοινωνικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτά να γίνονται σεβαστά στις δημόσιες συμβάσεις. Διαφανείς λοιπόν δημόσιες συμβάσεις από πλευράς δικαίου. Αυτό αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση ώστε να υπάρξει ένα ισότιμο πεδίο ανταγωνισμού για την καταπολέμηση της ε, απάτης και της διαφθοράς. Η ευρωπαϊκή αγορά δημοσίων συμβάσεων είναι πιο ανοιχτή ανά τον κόσμο. Αγορά δημοσίων συμβάσεων και αυτό θα πρέπει κάποιοι μηχανισμοί δημοσίων συμβάσεων να ενισχυθούν. Θα πρέπει να εξασφαλιστεί λοιπόν η διαφάνεια και να υπάρχει δικαιοσύνη σε ό,τι αφορά την ε, δαπάνη δημοσίου χρήματος. Θα πρέπει επίσης ε, να υπάρχει προσανατολισμός προς τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για να μπορούν και αυτές να συμμετέχουν σε διεθνούς διαγωνισμούς ε, και να τους ανατίθενται συχνότερα συμβάσεις γιατί συχνά αντιμετωπίζουν διακρίσεις σε ό,τι αφορά την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, για τι δημόσιε συμβάσει, νομίζω ότι θα πρέπει να επικεντρωθούμε στι εξαιρέσει στο τμήμα 3 και δει το άρθρο 9 που αφορά συμβάσει που εκχωρούνται με βάση διεθνεί διαδικασίε. Σε ό,τι αφορά την ε, ανάθεση συμβάσεων ε, παραδείγματο χάρη στον των αχυδρομικών υπηρεσιών, θα πρέπει να επικεντρωθούμε σε θέματα όπως ε, οι συμβάσεις που ανατίθενται σε σχέση με τη μίσθωση ή την επαναπόληση σε τρίτους ή για θέματα που έχουν να κάνουν με την άμυνα και για συμβάσεις που ανατίθενται στο πλαίσιο διεθνών διαδικασιών ή συμβάσεις που ανατίθενται σε εταιρείε ή κοινοπραξίες που έχουν σχέση μεταξύ τους ή σε μέλη κάποιου μήλου μιας κοινοπραξίας. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Η Έμα Μακλάρκιν τώρα έχει το λόγο από την ομάδα ECR. Ευχαριστώ πολύ. Η σημασία των ε, μεταρρυθμίσεων στον τομέα δημοσίων συμβάσεων είναι κάτι πολύ σημαντικό. Ξέρουμε ότι το 9% του ΑΕΠ τη Ευρωπαϊκή Ένωση προέρχεται από δημόσιε εξαγορέ αγαθών και υπηρεσιών και ίσω ανέβει το ποσοστό αυτό. γιατί μπορούν οι ανταγωνιστικέ βιομηχανίε και η αγορά δημοσίων συμβάσεων να αυξηθούν και να δημιουργήσουν θέσει εργασία όταν χρειάζονται οικονομικά κίνητρα και ρεθίσματα. Γι' αυτό λοιπόν θα συνεργαστώ ε, και εγώ με του συναδέλφου για να μπορέσουμε να εξυγχρονίσουμε τι δημόσιε συμβάσει. Η ομάδα μα, η CR, από την αρχή ηγείται όλη αυτή τη προπαρασκευή τη μεταρρύθμιση τα τελευταία δυόμιση χρόνια και αντιλαμβανόμαστε πλήρω τη δυνατότητα που έχουμε να μεταρρυθμίσουμε την, τον τομέα των διαγωνισμών ώστε να μπορεί να πληρεί τις ε, απαραίτητες προϋποθέσεις. Σε ό,τι αφορά τώρα το κανονισμό, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να πλουστεύσουμε και να κάνουμε πιο ε, σαφείς ε, τις οδηγίες, γιατί υπάρχει κίνδυνος μη συμμόρφωσης ε, και αυτό οδήγησε σε περιορισμό της καινοτομίας. Πρέπει όμως να βοηθήσουμε να αναδυθούν νέες πρακτικές ε, στις δημόσιες συμβάσεις και να γίνουμε κι εμείς πιο αποτελεσματικοί. Συμφωνώ με τον εισηγητή ότι θα πρέπει να είμαστε και προσεκτικοί ώστε την τρέξη οικονομική κατάσταση να μην τη χρησιμοποιήσουμε ως πρόσχημα για προστατευτικά μέτρα και λιγότερη διαφάνεια στην όλη διαδικασία. Τέλος, πιστεύω ότι είναι ευκαιρία και εμείς να προσαρμόσουμε τους κανόνες μας στην ψηφιακή εποχή ώστε οι δημόσιες συμβάσεις να συμβάλλουν με τη σειρά τους στην τόσο αναγκαία ανάπτυξη. Εμείς θα συνεργαστούμε ε, με όλους τις διάφορες επιτροπές. Ελπίζω να παραμείνουμε στο προσκήνιο και στην πρώτη γραμμή των μεταρρυθμίσεων γιατί είναι προτεραιότητά μας και η Επιτροπή μας ε, συγκεκριμένα ε, θα έχει και αυτή ένα πολύ σημαντικό ρόλο και ελπίζω και εγώ να συμμετάσχω ενεργά. Ο Γιάννη Ζαντό έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πράγματι πρόκειται για ένα εξαιρετικά σημαντικό θέμα δημόσιες ε, αγορές σε μια κατάσταση όπου τα μέσα είναι πενιχρά, όπου το εμπόριο δεν είναι απελευθερωμένο, οι δημόσιες αγορές θα πρέπει να αποβούν ένα εργαλείο στην υπηρεσία των οικονομιών μας. Και καταλαβαίνω τα όσα λέγονται για την αμοιβαιότητα και κάτι την θεμητό. Το ερώτημα το οποίο θα πρέπει να θέσουμε εξίσου είναι σε ποιο βαθμό οι δημόσιες συμβάσεις ε, μπορούν να αποβούν επίσης ένα εργαλείο στην υπηρεσία των επιχειρήσεών μας και ε, προστασία ε, ενός, τμήματος, ενός μέρους των επιχειρήσεών μας σε ένα τομέα που μπορούμε να θεωρήσουμε ότι έχει στρατηγική σημασία. Για παράδειγμα, η Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα συμμετέχει σε μια σύγκρουση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Καναδά για την ενεργειακή πολιτική η οποία ευνοεί τις ε, ντόπιε επιχειρήσεις όταν το ζητούμενο είναι να απτυχθούν ε, πράσινες τεχνολογίες. Για μένα κάτι είναι το αντίστροφο αυτό που θα πρέπει να γίνει. Σήμερα, για παράδειγμα, αυτός ο τομέας της ε, πράσινης ενέργειας είναι ένα τομέα που έχει μια εξόχω ε, στρατηγική σημασία και αν ε, η Κίνα έχει ένα πλεόνασμα παραγωγής φωτοβολταϊκών, είναι όπως όταν είχε ε, ε, ε, προσπαθώντας να σκοτώσει ολόκληρη την βιομηχανία, την παγκόσμια βιομηχανία φωτοβολταϊκών και 85% είναι, από την Κίνα. Και βλέπουμε ότι άλλες χώρες αντιδρούν. Οι βιομηχανίες ε, εξαφανίζονται, συρρυκνώνονται στην Ευρώπη και στην Αμερική και θα, η μόνη που θα επιβιώσει στην αγορά θα είναι οι Κινέζοι. Εγώ δεν έχω τίποτα κατά της Κίνας, αλλά το θέμα μου είναι ότι σε ένα τέτοιο τομέα κλειδί ε, θα πρέπει να επιχειρήσεις στη δική μας επικράτεια ε, ασκούν μια πολιτική, να μια για την ανανεώσιμη ενέργεια. Ε, για μένα πρόκειται για ένα ουσιώδες διακύβευμα που δεν μπορούμε να το επιλύσουμε αποκλειστικά ε, με τεχνικές προδιαγραφές. Μπορούμε βεβαίως με αυτό το μέσο να παρακάμψουμε το άνοιγμα της αγοράς των δημοσίων συμβάσεων για να ευνοήσουμε ορισμένους τύπους βιομηχανιών, αλλά δεν αρκεί. Ε, θα πρέπει από πολιτική άποψη αυτό που αφορά τις δημόσιες δαπάνες να μπορεί να ευνοεί επιχειρήσεις στη δική μας επικράτεια, την ευρωπαϊκή. Και θεωρώ ότι αυτό είναι πραγματικά ουσιώδες, γιατί αυτή η συζήτηση έχει, υπάρχει ήδη στις χώρες μας, αλλά μέχρι στιγμής η ευρωπαϊκή ε, θέση δεν ε, λαμβάνει παρκώς υπόψη της αυτό το διακύβευμα. Τώρα, όσον αφορά τα κοινωνικά ζητήματα και τα θέματα του περιβάλλοντος, θα πρέπει να μπορούμε να λάβουμε υπόψη μας τον κύκλο ζωής των προϊόντων και να εσωματώσουμε, όπως είπε, το ζήτημα των υπεργολάβων, της υπεργολαβίας. Και βεβαίως θα πρέπει να εξασφαλίσουμε να υπάρχουν ε, ε, κάποιοι ε, αντικειμενικοί στόχοι σε σχέση με τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές πτυχές για να μην υπάρχουν αμφισημίες όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις και τις δημόσιες αγορές. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Έχω τέσσερα ερωτήματα προς την Επιτροπή. Το πρώτο ερώτημα αφορά λίγο το τομέα του Ζαν Λικουζαντό. Στην έκθεση της βιομηχανικής πολιτικής που ενέκρινε το Κοινοβούλιο αποφασίσαμε οι δημόσιες συμβάσεις να συνιστούν σημαντικό πυλώνα για την υποστήριξη της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και προτείναμε να υπάρχουν αντίστοιχες ποσοστώσεις για καινοτόμα προϊόντα όπως στις Ηνωμένε Πολιτείε ή στην Ιαπωνία και να θεσπιστεί κάτι τέτοιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, εάν ε, δεν θεωρείτε ότι να αφιβόλω μια τέτοιου είδου ε, προσέγγιση για τη βιομηχανική πολιτική. Δεύτερον, πόσο σίγουρα είναι, βέβαια είναι η πρόταση ότι το κοινωνικό dumping και το περιβαλλοντικό dumping ε, εφαρμόζεται μέσω ε, λόγω προϊόντων που προέρχονται από τρίτες χώρες. Νομίζω ότι θα πρέπει να εξασφαλίσουμε στις ε, διμερείς εμπορικές συμφωνίες προϊόντα και υπηρεσίες που δεν παράγονται σύμφωνα με τους διεθνείς ε, κανόνες του ΑΕΛΟ να μην μπορούν να φτάνουν ε, μέσω του, της οδού των δημοσίων συμβάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τρίτον, ε, προσπαθούμε να ενισχύσουμε συστήματα θεμητού εμπορίου και να τα προωθήσουμε. Νομίζω ότι στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων θα πρέπει να εξασφαλίσουμε η ενίσχυση και η προώθηση του θεμητού εμπορίου να ενισχύει μικρούς παραγωγούς σε τρίτες χώρες. Αλλά κάτι τέτοιο δεν βλέπω να αναφέρεται στη δική σας πρόταση. Δεν ξέρω, σας απατώμε. Τέταρτον, όσον αφορά την οδηγία για τις συμβάσεις παραχώρησης. Εδώ ε, βρισκόμαστε στον ε, τομέα της δημόσιας πρόνοιας, όπου παραχωρούνται κάποιες συμβάσεις ε, στον τομέα του ύδατος, και άλλους τομείς. Είναι βέβαιο ότι οι συμβάσεις παραχώρησης μέσω των ε, κοινοτήτων μπορεί να παραμείνει ως έχει και να εξασφαλίζεται από τους Δήμους και τις κοινότητες ή θα ανοίξουμε το δρόμο για ανάθεση σε τρίτους. συντομία, κύριε Πρόεδρε, με ε, άρχισα να σηκώ όταν άκουγα για να τίθεται θέματα προστατευτισμού στι δημόσιε συμβάσει. Θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Είδαμε τι έγινε στην Αμερική και είδαμε τι έγινε στην Αργεντινή επίση ε, ε, πρόσφατα για προϊόντα που έρχονται από τρίτες χώρες. νομίζω ότι πρόκειται εδώ για τα χρήματα των φορολογουμένων. Άρα λοιπόν, εάν δημιουργήσετε μια κατάσταση όπου γίνεται μια παρέμβαση στην αγορά ε, μέσω επικοινοτρόπος ε, δεν παίρνετε την αξία των χρημάτων σας. Για παράδειγμα, στην, ε, στη Μεγάλη Βρετανία, για μια εταιρεία η οποία δεν, δεν μπόρεσε να της ανταθεί με δημόσια σύμβαση και τελικά πήγε στην Γερμανία. Αυτή είναι μια δεν ξέρω για αν μιλούσε για τον προστατευσμό. Δεν ξέρω γιατί μιλούσε ακριβώ. Τι, γιατί μιλούσε, Μιλούσες για μια ανοιχτή ελεύθερη αγορά. Δεν ξέρω. Και θα ήθελα να ακούσω ποια είναι η γνώμη της Κομισιόν. Thank ακούσουμε τώρα την Επιτροπή. Τρία ονόματα έχουν μπροστά μου. Mr. or Mrs. Ε, I'm not sure. Who Ποιος θα μιλήσει από την Επιτροπή. Σας παρακαλώ. Μιλήστε. Ποιος είναι τέλος πάντων υπεύθυνο. Uh, ε, um, ε, first of all, I'm, I'm afraid my name εγώ έχω να κάνω με το φάκελο που έχει να κάνει με, την παραχω... με τις και θα απαντήσω στο ερώτημα του κύριου Λάγκη. Αλλά πριν το απαντήσω το ερώτημα θέλω να μου το επαναλάβει, γιατί δεν το κατάλαβα πολύ καλά. Ε, what was the question about? If you, would kindly... Σας παρακαλώ λοιπόν να επαναλάβετε το ερώτημά σας. Im Moment äh, werden Konzessionen ja gerade von αυτή τη στιγμή ε, εκχωρούνται, παραχωρούνται κάποιες συμβάσεις από τους Δήμους και τις κοινότητες για διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Για παράδειγμα τα νοσοκομιακά ή η παροχή ύδατος. Και υπάρχουν ε, βεβαίως αποκλειστικά δικαιώματα για ορισμένους ε, παρόχους, αλλά υπό τον όρο να μην ε, δίδονται δημόσια κονδύλια για αυτές τις υπηρεσίες. Θα παραμείνει το κοθεστώς αυτό ως έχει ή τι θα γίνει, ε, θα υπάρξουν πάροχοι από τρίτες χώρες που θα εισδύσουν σε αυτό το τομέα τελικά των συμβάσεων παραχώρησης για δημόσιες υπηρεσίες. Yes, so um, I think that uh, uh, Κοιτάξτε, το πιο σημαντικό σημείο είναι να τονίσουμε πως η πρόταση για την οδηγία για τις ε, παραχωρήσεις αδειών δεν, είναι για την, δεν αφορά την ιδιωτικοποίηση ή την εξωτερική ανάθεση υπηρεσιών. Εάν σήμερα οι κοινοφιλείς υπηρεσίες τις οποίες αναφερθήκατε άμεσα προσφέρονται από τις κοινοτικέ υπηρεσίες από τους ίδιους πόρους τους, η πρόταση δεν αμφισβητεί αυτή την κατάσταση. Δεν υπάρχει υποχρέωση για εξωτερική ανάθεση που να προκύπτει ή να απορρέει από τις διατάξεις της οδηγίας. Ομοίως, αν κάποιος Δήμος ε, επιθυμεί να παρέχει αυτές τις υπηρεσίες μέσω ενός φορέα εντός του Δήμου, δεν μπορεί να το κάνει και μάλιστα θα έλεγα ότι αυτή η δυνατότητα ενισχύεται μέσω του καθορισμού των όρων περί Εσωτερική προσφορά ή παροχή των υπηρεσιών αυτή. Πρώτα δεν αλλάζει λοιπόν τίποτα εκεί. Αν όμω υπάρχει απόφαση ενό Δήμου για εξωτερική ανάθεση αυτών των υπηρεσιών σε τρίτου, δημόσιους ή δηλαδή που δεν είναι εσωτερική αλλά είναι δημόσιες φορές ή δημόσιοι φορείς ή ιδιωτικοί φορείς, εκεί Ήδη ε, επί τη βάση των αρχών της συνθήκης δεν μπορούν να αναθέσουν τέτοιες, ε, την παροχή αυτών των υπηρεσιών άμεσα. Και αν αυτή η οδηγία τελικά εγκριθεί, οι Δήμοι θα οφείλουν να ακολουθούν κάποια διαδικασία και να τηρούν κάποιους κανόνες ε, ώστε να αναθέσουν αυτές τις παραχωρήσεις. Πάντως, δεν θα έχει αυτό επίπτωση για το αν θα πρέπει ή όχι άμεσα το κράτος να παρέχει την συγκεκριμένη υπηρεσία ή αν θα πρέπει ε, ε, να την αναθέσει σε τρίτο φορέα. Επίσης, να τελειολοκληρώσω με τη διεθνή πτυχή, να θυμίσω πως αυτή τη στιγμή οι παραχωρήσεις δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε, οποιαδήποτε διεθνή όπω όπως η GPA, η υποψήφια από τρίτες χώρες ή από ε, του ε, GPA θα βρίσκονται στην ίδια θέση όπως και οι υποψήφοι στις, ε, για δημόσιες συμβάσεις που δεν προέρχονται από χώρες GPA. Any other contribution from the Commission? Κάποιος άλλο από την Κομισιόν θέλει να πάρει το λόγο. Μάλιστα κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου να σας παρουσιαστώ γιατί έχετε ένα κατάλογο. Ονομάζομαι Νάντια Κώστα Κόρτα και εδώ αντιπροσωπεύω τις υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Εξωτερικής Αγοράς που είναι αρμόδιες για τη μεταρρύθμιση την ίδια των δημοσίων συμβάσεων. Εγώ θέλω να απαντήσω στην ερώτηση του κυρίου Λάγκια αν κατάλαβα καλά όσον αφορά τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Πρόκειται για ανησυχία, για της Κομισιόν που θέλει να αποφύγει στο πλαίσιο των δημόσιων συμβάσεων να γίνουν δεκτές προσφορές ε, ε, ετών, ετούντων που δεν σέβονται τις διατάξεις ε, τις κοινωνικές και τις περιβαλλοντικές και η Κομισιόν στις προτάσεις της έχει προβλέψει ακριβώς έτσι ώστε να καταπολεμήσει το κοινωνικό και περιβαλλοντικό ντάμπινγκ διάφορες διατάξεις που συνίστανται στη δυνατότητα να εξαιρούνται οι προσφορές που δεν τηρούν αυτούς τους όρους. Είναι δυνατόν, αλλά αυτό δεν είναι υποχρέωση της συμβαλόμενης αρχής να μην, χωρίσει, να μην συνάψει σύμβαση με κάποιον οικονομικό φορέα του οποίου η προσφορά δεν σέβεται τις υποχρεώσεις στον κοινωνικό τομέα, ας πούμε το δίκαιο το εργατικό ή το δίκαιο περί περιβάλλοντος, καθώς επίσης και όσον αφορά τις, κοινωνικές και, τις διεθνείς κοινωνικές και περιβαλλοντικές διατάξεις που απαριθμώνται σε ένα προσάρτημα στην πρόταση οδηγίας. Υπάρχει δηλαδή δυνατότητα απόρριψης της προσφοράς. Επίσης προβλέπεται οι συμβαλόμενες αρχές να μπορούν να αποκλείσουν οικονομικούς φορείς όταν οι συμβαλόμενες αρχές γνωρίζουν πως ο συγκεκριμένος οικονομικός φορέας έχει παραβιάσει αυτές τις ίδιες υποχρεώσεις, τις ευρωπαϊκές ή τις διεθνείς. Εκεί λοιπόν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας εξ αρχής και όχι η προσφορά του. Τρίτη πτυχή στην πρόταση της Κομισιόν είναι αυτή που αφορά τις ε, φύσικα χαμηλές προσφορές. Εδώ πρόκειται για μια υποχρέωση, υποχρέωση της συμβαλόμενης αρχής να αποκλείσει τις προσφορές όταν βλέπουμε ότι λόγω προσφορές είναι φυσικά χαμηλές λόγω παραβίασης ευρωπαϊκών ή διεθνών υποχρεώσεων ε, στον κοινωνικό και περιβαλλοντικό τομέα. Ελπίζω έτσι να απάντησα στο ερώτημά σας και θα ήθελα να δώσω το λόγο και στον συνάδελφο Βόλμαν, ο οποίος ε, ασχολείται πιο συγκεκριμένα με τις, το, το διεθνές επίπεδο. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο σε σχέση με τον κανονισμό ο οποίος εγκρίθηκε την 21η Μαρτίου για την πρόσβαση τρίτων χωρών ε, στην ε, αγορά δημοσίων συμβάσεων τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, δεν είναι στην μέση διάταξη άμεση αυτό το θέμα, αλλά πολλέ ερωτήσει είχαν να κάνουν με αυτό το νέο μέσο και γι' αυτό θα ήθελα να κάνω κάποιε διευκρινήσει. Πρώτα απ' όλα, Φυσικά η Ευρωπαϊκή Ένωση βιώνει μια χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση. Κατά την άποψή μας λοιπόν είναι σημαντικό σε αυτό το πλαίσιο να έχουμε και μέσω των δημοσίων συμβάσεων την βέλτιστη δυνατότητα, τη βέλτιστη μάλλον σχέση τιμής και αποτελέσματος. Έχουμε την ε, συμφωνία GPA για τις ε, ε, δημοσίες συμβάσεις είμαστε ανοιχτοί, ε, η αγορά δηλαδή τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ανοιχτή σε όλου του τομεί, αλλά αν θέλουμε να έχουμε πρόσβαση σε τρίτε χώρε. βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι αντιμετωπίζουμε πρόβλημα, δεν μπορούμε να έχουμε επαρκή πρόσβαση αγορά σε τρίτες χώρε. Εξού πιστεύουμε ότι είναι απαραίτητο να δημιουργηθεί ένα μέσο το οποίο θα μας δώσει τη δυνατότητα να ασκήσουμε μόχλευση απέναντι σε τρίτες χώρες και έτσι θα μπορούμε να διαπραγματευτούμε ένα μεγαλύτερο μερίδιο στην αγορά, πρόσβαση καλύτερη στην αγορά σε κάποια στιγμή. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μία διάταξη για την πρόσβαση τρίτων χωρών, ε, το άρθρο 58 δηλαδή της οδηγίας ε, για τις κοινοφιλείς υπηρεσίε, αλλά τίποτα άλλο. Άρα λείπει εντελώ ε, μια εξωτερική πολιτική διαγωνισμών, να συμβάσω. Τώρα, σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο τη πρόταση, Υπήρξε διαίρεση των ε, μπλεκομένων σε σχέση με την πρόταση. Οι εταιρείε ήθελαν να κλείσει η αγορά, οι δημόσιε αρχέ εν γέννη ήθελαν να παραμείνει η σημερινή κατάσταση. Η Κομισιόν ακολούθησε τη μέση οδό. Δηλαδή, λίγο πολύ λέμε ότι βασικό ε, κανόνα τη ε, αγορά των δημόσιων συμβάσεων είναι το άνοιγμα. Μόνο αν υπάρχει πρόβλημα θα μπορεί να θέσει αρχέ να εξηγεί, ε, να ε, εξαιρέσουν, να αποκλείσουν κάποια ξένα τμήματα και να κλείσουν ένα συγκεκριμένο ε, στοχευμένο κομμάτι της αγοράς δημοσίων της Μέσης Ένωσης. Αυτός είναι ο βασικός κανόνας περιλαμβάνει αυτό το μέσο. Αργότερα φαντάζομαι ότι θα γίνουν μεγαλύτερες συζητήσεις για αυτό το μέσο, αλλά αυτή είναι η πρώτη γενική επισκόπηση. Ναι, πράγματι δεν είναι ακόμα στην ημερησία διάταξη. Ο Γιάννη Ξαντό, θέλει κάτι να ρωτήσει. Ναι, για το τοπικό περιεχόμενο θέλω μια απάντηση παρακαλώ. Ναι, πράγματι ήταν ένα ερώτημα προς την Κομισιόν. Για το δημόσιο περιεχόμενο. Όπως σας είπα, ο βασικός κανόνας είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ανοιχτή και υπό ορισμένες συνθήκες μπορεί να αποκλειστεί διαγωνισμός όταν μια χώρα διαθέτει υπηρεσίε ή ε, που δεν εμπίπτουν, ε, που δεν τηρούν τις ε, προποθέσει Ευρωπαϊκή Ένωση. Απάντησε το ερώτημά σα. Όχι. Τέλο πάντων, Α πάμε πάλι στον Τζαν Λούκα Σούστα για να κλείσει. Σα ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να σας θυμίσω ότι η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών είναι 25 Ιουνίου και ότι 20 και 21 Ιουνίου θα ε, συζητήσουμε την έκθεση. Η συζήτηση ήταν πολύ ζωντανή και πολύ ενδιαφέρουσα και εξάλλου το θέμα είναι ουσιώδες. Γνωρίζουμε ότι μέγα μέρος της ανάκαμψής μας και της ανταγωνιστικότητάς μας εξαρτάται από την αναδιοργάνωση της εσωτερικής αγοράς και αγοράς των δημοσίων προμηθειών των δημοσίων συμβάσεων είναι πολύ σημαντικός. Ε, πιστεύω και από τις τροπολογίες που θα υποβάλουμε και εγώ ίδιος αλλά και οι συνάδελφοι της ομάδας μου αλλά και των άλλων ομάδων θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τη δική μας ιδιαίτερη θεσμική θέση που είναι ή που θα έπρεπε να βασίζεται κυρίως σε κριτήρια επικουρικότητας. Υπάρχουν ζητήματα όπως αυτά που ανέφερε ο συνάδελφος Ζαντό που είναι χαρακτηριστικές για μια τοπική διάσταση, μια ισχυρή σχέση ανάμεσα στην κοινότητα, την ε, επικράτη και την παραγωγική δυνατότητα και που κατά κάποιο τρόπο θα πρέπει να διατηρηθούν. Ας πούμε, ας πούμε τη διοργάνωση των υπηρεσιών για τα, τις καντίνες των σχολείων και άλλου είδους τέτοια πράγματα, τα οποία δεν μπορούμε να αφήσουμε ε, να ρυθμιστούν σε διεθνές επίπεδο. Αναφίβολα κάποιες αρχές που περιλαμβάνονται στις προτάσεις της Κομισιόν ε, σχετίζονται και πάλι με μια παραχώρηση, εκχώρηση που είναι χαρακτηριστική του φιλελευθερισμού που ήταν χαρακτηριστικός εδώ και λίγα χρόνια. Εντάξει να ανοίξουμε την αγορά, αλλά μέσα σε ένα πλαίσιο το οποίο να σέβεται την επικουρικότητα. Δηλαδή υπάρχουν βασικά θέματα που αφορούν τις, τα έργα υποδομής, τις μεγάλες σχέσεις με τον κόσμο, τις μεγάλες, τους μεγάλους ε, διαγωνισμούς όπου εμείς συζητάμε αμοιβαιότητα στις διεθνείς αγορές. Υπάρχουν άλλα θέματα που αφορούν την εγκύτητα και εκεί θα πρέπει να προβλέψουμε αποκλειστικότητα ή τη δυνατότητα αποκλειστικότητας, ούτως ώστε οι τοπικές ε, πραγματοκα... Ε, ε, αρχές να μπορούν να ρυθμίσουν τα πάντα. Να μην ξεχνάμε την οδηγία Μπόλκενστάιν, και τα μειονεκτήματά της, αλλά να μην δημιουργήσουμε και προϋποθέσεις για μια, ένα υπερβολικό κλείσιμο που θα φρενάριζε τις δυνατότητες της ενίας αγοράς. Να είναι στο πρωτοπορία η Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τις αρχές που χαρακτηρίζουν την ίδια της ε, θεσμική διάσταση. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Πολύ μεγάλη πολιτική σημασία η έκθεση αυτή. Η συζήτηση του σχεδίου έκθεσης θα είναι τον Ιούνιο σε δύο μήνες και προβλέπεται η ψηφοφορία για το Σεπτέμβριο. Έχουμε μπόλικο χρόνο λοιπόν για να σκεφτούμε όλο αυτό το πακέτο. 22. Σημείο 22. The so-called market access. Κανονισμός περί πρόσβασης στην αγορά. Κανονισμός του 2007 που επέκτηνε τις μονομερείς προτιμήσεις για τις χώρες ΑΚΕ που διαπραγματεύονται τις ε, ε, συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης. Πρόκειται για νομοθετικό θέμα. Εμείς είμαστε οι αρμόδιοι από τις ουσίες επιτροπής. Η μας είναι ο David Μάρτιν. Ήδη έχει γίνει μια ανταλλαγή απόψεων και τώρα εξετάζουμε το σχέδιο έκθεσης του εισηγητή που το έχετε στους φακέλους σας. Και δίνω το λόγο στον εισηγητή David Μάρτιν. Ε, από την ομάδα του Σοσιαλιστών. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομο γιατί, όπω είπατε, το έχουμε ξανασυζητήσει το θέμα. Αλλά, καθώ είπατε κιόλα, είναι από τμήμα του πακέτου των συνεχιζόμενων διαπραγματεύσεων σε σχέση με τις ε, συμφωνίες ε, οικονομικής εταιρικής σχέση, Όπως ξέρετε, η εξαίρεση του ΠΟΕ ξέπνευσε τον Ιανουάριο του 2007. Τότε για να μπορέσουμε να τηρήσουμε την προθεσμία. Θα θυμάστε, συνάδελφοι, ότι αρκετές χώρε ξεκίνησαν ε, τέτοιε οικονομικές συμφωνίες, εταιρικέ σχέσεις και μάλιστα ορισμένες χώρες καραβικές ε, συνήψαν, συνήψαν ε, πλήρεις συμφωνίες τέτοιου τύπου. Οι διαπραγματεύσεις με πολλές αφρικανικές χώρες δεν ήταν ε, τόσο <laughs> ταχύες και μας απογοήτευσαν. Σε κάποιες περιπτώσεις δεν καταφέραμε καν να διαπραγματευτούμε, σε άλλες κάναμε κάποιες αρχικές συμφωνίες οι οποίες δεν έχουν εφαρμοστεί, έχουν μονογραφεί αλλά δεν έχουν επικυρωθεί και ούτω καθεξής. Εάν είχε εκπνεύσει η εξαίρεση του ΠΟΕ χωρίς να υπάρξει κάποια πρόβλεψη. Πολλές χώρες θα έμεναν εκτός της αγοράς μας. Ε, γι' αυτό και καλύψαμε αυτό το κενό μέσω αυτού του κανονισμού που είναι ο κανονισμός περί πρόσβασης στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης έτσι ώστε 26 χώρες από αυτές που συμπεριλαμβάνονταν στην εξαίρεση του ΠΟΕ να συνεχίσουν να έχουν πρόσβαση στην αγορά μας. Η πρόταση της Κομισιόν είναι ότι ήγηκε πλέον η ώρα να πάψει να ισχύει αυτός ο κανονισμός και να οριστεί η ημερομηνία της 1ης Ιανουαρίου 2014 οπότε και θα πρέπει να επικυρωθούν οι συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης ή αλλιώς οι χώρες που δεν θα το έχουν κάνει αυτό να επανέλθουν στο καθεστώς γενικών προτιμήσεων ή εν πάση περιπτώσει να ε, ε, δεχτούν τις συνέπειες. Οι χώρες όμως που θα χτυπηθούν περισσότερο θα είναι η Μποτσουάνα και η Ναμίμπια, που δεν θα έχουν καν για συμφωνία γενικευμένων προτιμήσεων, γιατί δεν είχαν πριν. Έχουμε και την συμφωνία όλα εκτός από όπλα και θα βρεθούν σε ανταγωνιστικό μειονέκτημα προσπαθώντας να έχουν πρόσβαση στην αγορά μας. Επισκεφθήκαμε μαζί με άλλα δυο μέλη της Επιτροπής μας στην Κένια που εξέφρασε μεγάλες ανησυχίες όσον αφορά την εκπνοή του κανονισμού για την πρόσβαση στην αγορά, ιδιαίτερα για την βιομηχανία ανθών που θα αντιμετωπίσει 24% μείωση, συρρήκνωση, αν δεν έχει γίνει δεν έχει ολοκληρωθεί η διαπραγμάτευση της οικονομικής εταιρικής σχέσης. Θα έχει αυτό μεγάλο αντίκτυπο στην οικονομία. Τι να κάνουμε λοιπόν. Από τη μια άλλη πλευρά δέχομαι τη λογική της Κομισιόν ότι πρόκειται για προσωρινή λύση και ότι κάποια στιγμή η προσωρινή λύση θα πρέπει να πάψει να λειτουργεί. Χωρίς την εξαίρεση θα ε, ε, βρισκόμασταν σε παραβίαση των κανονισμών του ΠΟΕ. Και αν αυτή η, αυτός ο κανονισμός συνεχίζει να ισχύει, πάλι θα ε, ε, είναι σαν να παραβιάζουμε τους κανόνες του ΠΟΕ. Χρειάζεται μια καταληκτήριος προθεσμία. Το ερώτημα λοιπόν δεν είναι αν χρειάζεται ε, ημερομηνία λήξη, αλλά το πότε θα είναι αυτή. Η Κομισιόν προτείνει το 2014, τον Ιανουάριο του 2014. Εγώ νομίζω πω είναι πολύ σύντομα και μιλώντα με του εταίρου μας των χωρών ΑΚΕ, Κανένα δεν χρησιμοποίησε τη λέξη εκβιασμό, αλλά πολλοί θεωρούν ότι είναι πολύ ε, μεγάλη πίεση να του αναγκάσουμε να υπογράψουν αυτέ τι συμφωνιε τόσο σύντομα, βιαστικά, βιαστικά. Εγώ προτείνω να υπάρξει μια προθεσμία δύο χρόνια αργότερα, δηλαδή 1η Ιανουαρίου 2016. Να σα δώσω ένα παράδειγμα. Η Κένια μπορεί, αν τα καταφέρει, να υπογράψει μια ε, συμφωνία Ιούνιο-Ιούλιο. Αν όχι, περνά σε ένα φθινόπορο προεκλογική εκστρατεία, εκεί δεν θα συμβεί τίποτα. Μετά θα είναι η μεταεκλογική εκστρατεία που θα σχηματιστεί η κυβέρνηση και μετά θα πρέπει να ξαναρχίσουν διαπραγματεύσει και θα έχει φτάσει 1η ε, Ιανουαρίου 2014. Θα ήταν άδικο. Αν πάμε στις άλλες δύο χώρες, Μποτζουάνα και Ναμίμπια, οι περισσότεροι φοβούνται ότι το πρόβλημα που έχουν αυτές οι χώρες δεν είναι ε, δικό τους, δεν είναι το πρόβλημα εκείνων. Θα ήταν σχετικά εύκολο για αυτούς να πούνε ναι στην συμφωνία αυτή, η δυσκολία που έχουν με την Νότια Αφρική. Αυτό τους εμποδίζει να ε, συνυπογράψουν αυτή τη συμφωνία και άρα χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να βρουν λύση με τους γείτονές τους. 2016. Πρώτη, ε, πρώτου 2016 λοιπόν. Δεν μπορεί να αφαιθεί ανοιχτή η λήξη. Μάλιστα. Σολομόντιος πρόταση. Ας περάσουμε στη συζήτηση. Σκιώδης, Σκιώδης και ο Κρίστοφερ Φιάλλαν έχει ζητήσει το λόγο από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σε ευχαριστούμε, Ντέιβιτ. Καταλαβαίνω πολλά πράγματα όταν ακούω τα όσα λέει ο Ντέιβιτ και τις ε, ανησυχίες που εκφράζει. Παρ' όλα αυτά, έχω κάποιες δυσκολίες να αποδεχτώ την επέκταση της ε, προθεσμίας και θα σας πω ποια, ποιοι είναι οι λόγοι μου. Καταρχήν, η διαπραγματεύσεις για τις συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης ξεκίνησαν το 2007. Δηλαδή έχουμε 7 χρόνια που είναι πολύς χρόνος. Ορισμένοι κατέληξαν και συνήψαν τις συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης και νομίζω ότι δεν είναι έντιμο απέναντί τους. Ε, γιατί στην περίπτωση αυτή ποια είναι τα κίνητρα που δίνουμε στους άλλους και τι μήνυμα θέλουμε να περάσουμε. Επίσης, τι πιστεύουμε ότι θα συμβεί, ποιες θα είναι οι συνέπειες. Δηλαδή θα δώσουμε κάποιον έξτρα χρόνο κατ' ουσία θα αποδυναμώσουμε τη βούληση να συνάψουμε τις ε, συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης ή τελικά θα ξυπνήσουμε τον χρόνο αυτό και θα καταλήξουμε μετά από αυτή την προθεσμία σε αυτές τις συμφωνίες. Και Νομίζω ότι είναι καλό στο πλαίσιο αυτό να δούμε τι γίνεται με συγκεκριμένες χώρες, για παράδειγμα την Κένια που αναφέρατε. Και πάντοτε όταν κάνουμε τις συζητήσεις τελικά καταλήγουμε ότι σε μια χώρα επίκυνται εκλογές. Και τελικά ε, εκπονούμε τα χρονοδιαγράμματα σε συνάρτηση με τις εκλογές, τις ημερομηνίες των εκλογών. Αλλά στη συνέχεια βλέπουμε ότι γίνονται εκλογές και δεν αλλάζει τίποτα. Επίσης, είναι αλήθεια τόσα είπατε για την Ποτσβάνα και την Αμίμπια. Αλλά μπορούμε να βάλουμε δύο χρόνια. Αλλά και μετά τι θα γίνει με τη Νότια Αφρική. Και έχει νόημα να δώσουμε άλλα δύο χρόνια. Στο ΕΛΚ ε, θέλουμε μια πιο νομική προοπτική. Εγώ δεν είμαι νομικός εξ επαγγέλματος, αλλά ε, ε ίσως ε, ε, θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με το ισχύον καθεστώς. Η, επέκταση του, η χρονική του επέκταση ίσως δημιουργήσει κάποια επιπλέον προβλήματα και θέσει επιπλέον προκλήσεις. Άρα λοιπόν νομίζω ότι το ΕΛΚ θα συμφωνούσε με την πρόταση της υποτροπής. Δηλαδή, ίσως η τήρηση αυτού του χρονοδιαγράμματος των 7 ετών είναι αυτό που επιθυμούμε για την ολοκλήρωση αυτών των συμφωνιών, την οποία επιθυμούμε. Γιατί η λύση δεν μπορεί να είναι άλλη παρά η σύναψη μιας συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης. Πρόεδρος. Ο επόμενος σκιώδης είναι ο Νίκολα Ρινάλντι. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εγώ υποστηρίζω μια θέση που είναι υπέρ της πρότασης της Επιτροπής και της προθεσμίας που θέτει η Επιτροπή για αρκετούς ε, λόγους που χρειάζεται να τους επαναλάβουμε. Οι συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης δεν ξεκίνησαν το 2007, αλλά επρόκειτο να ολοκληρωθούν το 2007. Ξεκίνησαν κατ' ουσία το 2001. Έχετε δίκιο. Βρισκόμαστε, εξαντλούμε τον επιπλέον χρόνο. Έχουμε όλο επιπλέον κι άλλος και άλλος χρόνος. Δίδεται. Και εγώ, εμένα μου έκανε κάποια εντύπωση η συζήτηση στην Επιτροπή Ανάπτυξης, της οποίας είμαι μέλος, και οι οποίοι δεν θέλουν καμία προθεσμία. Ακόμα και η δική μου ομάδα όπως εκπροσωπείται εκεί. Για λόγους που σχετίζονται ακριβώς με την ανάπτυξη. Τώρα, τα όσα λέει ο Κρίστοφερ είναι απολύτως ορθά αλλά θα πρέπει να πω ότι συμφωνώ με την πιο σολομόντια προσέγγιση του εισηγητού. Μάλιστα. Γιατί δεν υπάρχει μια ιδανική κατάσταση. και δεν νομίζω ότι ε, μπορούμε να έχουμε μια επιλογή. Θα πρέπει να, θα πρέπει να κάνουμε μια επιλογή και θα πρέπει να πάρουμε τα συν και τα κατά της κάθε θέσης. Και υπό μία έννοια, το να λάβουμε υπόψη μας όλα τα διαφορετικά στοιχεία σε αυτή τη φάση, εάν θέλουμε να περιμένουμε άλλα δύο χρόνια και ενδεχομένως να καταλήξουμε σε μία συμφωνία ή να περιμένουμε άλλο ένα χρόνο, αυτό θα σημαίνει το τέλος της Συμφωνίας Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης. Και το γεγονός ότι βρισκόμαστε μέσω συνεχών παρατάσεων είναι ένα επιχείρημα του να πούμε αν αυτές οι χώρες χρειάζονται ένα-δύο χρόνια παραπάνω, ε, κάτι τέτοιο δεν θα είναι ολέθριο για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για, το, για τις ίδιες της Συμφωνίας Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης. Παρ' όλα αυτά θα ήθελα να θέσω δύο διευκρινιστικές ερωτήσεις. Η πρώτη, εάν δεν έχουμε μια προθεσμία θα έχουμε προβλήματα στον ΠΟΕ. Είμαστε ήδη σε μια κατάσταση όπου ενδεχομένω θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε προβλήματα στον ΠΟΕ. Εάν αναβάλουμε την οριστή σε ημερομηνία, David, αυτό είπε θα μπορούσε να προστατεύσει την Ευρωπαϊκή Ένωση από τυχόν αντιδράσει εντό του ΠΟΕ. Ε, κατανοώ το επιχείρημα ότι ναι μεν αναβάλουμε, παρατείνουμε, αλλά μετά θα πρέπει να δοθεί ένα τέλος. Αυτό θα μπορούσε να συνιστά ένα επιχείρημα στη Γενέβη, αλλά θα πρέπει να μα δώσει κάποιες διευκρινήσει ε, εφόσον τις διαθέτεις. Δεύτερον, γιατί μιλάμε, γιατί όγκους ε, εμπορίου μιλάμε, έχουμε καθόλου στοιχεία, γιατί εν γέννη οι συμφωνίες ε, Ευρωπαϊκή Ένωση ΑΚΕ είναι ισχνές σε σχέση με το παγκόσμιο όγκο εμπορίου και τελικά θα δημιουργήσουμε περισσότερα προβλήματα. Ο Ευχαριστώ πολύ κύριε ε, Πρόεδρε. Συμφωνώ με τον Κρίστεφερ. Το πρόβλημα, David, είναι ο κύριο. Στέρντι. Ε, εδώ θα διαφωνήσει μαζί μου, αλλά Επιτροπή την εποχή εκείνη ε, ήθελε να επιβάλλει τους όρους τους και δημιούργησε ένα νέο πνεύμα το οποίο παραμένει και το οποίο δημιούργησε όλα αυτά τα προβλήματα κατά την άποψή μου. Αλλά αν δεν θέτουμε κάποια ημερομηνία και δεν τη τηρούμε, θα θέλουν συνεχώς να παρατείνουν την ημερομηνία και αυτό δεν είναι έντιμο σε σχέση με εκείνους που ήδη υπέγραψαν και ανταπεξήλθαν σε όλες αυτές τις ισχυρές διαπραγματεύσεις. Δεν είμαι σίγουρος λοιπόν ότι συμφωνώ μαζί σου όσον αφορά την παράταση της προθεσμίας. Και το άλλο θέμα εδώ για την αναβολή είναι ότι ε, ε, υποθέτεις ότι θα επανεκλεγείς και ότι θα ξανά είσαι εισηγητής. Ισχύει όμως αυτό. Και ώρα από τους Πρασίνους. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, να ευχαριστήσω Σαν για την εκθεσή του. Πρέπει να πω ότι είχαμε συνδυάσει στο Στρασβούργο, η Σκιώδης και ο κύριος Μάρτιν, και εγώ είχα πει ότι ο Ντέιβιτ έδειχνε ότι δέχεται τα σημεία τα οποία εμείς ε, σχολιάζαμε, δηλαδή ότι ζούμε σε έναν κόσμο που δεν είναι τέλειος και ότι αν κάθε χώρα και είχε, ήθελε μια τέτοια συμφωνία, τότε θα ήταν τέλειος ο κόσμος. Υπάρχει ε, μια πίεση στις χώρες ΑΚΕ, η οποία είναι δυσανάλογη με την οικονομική αξία. είτε δεν είναι ε, διατεθειμένες να πάνε προς αυτή την κατεύθυνση, είτε δεν μπορούν δεν έχουν την υποδομή. Και το Συμβούλιο Υπουργών το 2011 τον χρόνο και είχε πει ότι οι κανονισμοί θα μεταφέρουν, θα μετατοπίσουν ακόμη περισσότερο κέντρο βάρος ε, και μάλιστα εις βάρος των χωρών και, και γι' αυτό και το απέρριψαν αυτό οι αρχικές χώρες και όταν πιέζονται νιώθουν ότι είναι υποχρεωμένε ουσιαστικά να συνάψουν τέτοια συμφωνία οικονομική εταιρική σχέση. Εμείς δεν δεχόμαστε τα επιχειρήματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπέρ του κανονισμού. Δεν είναι βάσιμα. Δεν αληθεύει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συρθεί ενώπιον του ΠΟΕ εάν δεν εγκριθεί ο κανονισμός. Πολύ λίγες είναι αυτές οι ε, πιθανότητες να κινήσει δηλαδή η διαδικασία οποιαδήποτε χώρα. Και το σύστημα κινητικών προτιμήσεων, το GSP, δεν είναι εναλλακτική λύση. Υπάρχουν πολλά ε, προϊόντα, προκυπευτικά, κακάο κτλ. που θεωρούνται ευαίσθητα. Δεν θα εντάσσονταν λοιπόν στις διευθετήσεις ε, GSP. Και το πρώτο τελευταίο μου σημείο. Μας εκπλήσει η IT που ξέρουμε ότι έχει πληγεί από τεράστιους ε, τυφώνες πριν από δύο χρόνια, να μπαίνει στις χώρες που απειλούνται με την απόσυρση ε, αυτών των προτιμήσεων εάν δεν υπογράψει Συμφωνία Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης. Ο Ντέιβιτ ε, έχει υποσχεθεί ότι θα προτείνει αναβολή της ε, έναρξης ισχύω του κανονισμού για μια ακόμα διετία. Εγώ όμως νομίζω ότι η κατάσταση θα είναι η ίδια και τότε. Γι' αυτό σας παρακαλώ να αναθεωρήσετε την έκθεση σας κύριε Μάρτιν και να συστήσετε τελικά απόρριψη του κανονισμού. Πρόεδρος, επιτρέψατε μου να κάνω και εγώ μια παρατήρηση. Υπάρχει πάντα το έρμπας και πάντα θα υπάρχει όφελος. Κύριος Λάγκια από τους Σοσιαλιστές τώρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, νομίζω ότι θα πρέπει όλοι να ομολογήσουμε ότι οι διαπραγματεύσεις για τη Συμφωνία Οικονομικών Εταιρικών Σχέσεων δεν έχουν μόνο αποτύχει επειδή δεν έχουν συμμορφωθεί οι εταίροι μας, αλλά και επειδή η Ευρωπαϊκή ε, Επιτροπή η οποία ε, ηγείται των διαπραγματεύσεων δεν ε, είχε τόσο εταιρική δομή. Λοιπόν, εάν πάρουμε σοβαρά το θέμα αυτό των εταιρικών σχέσεων, θα πρέπει να υπάρξει μια εταιρική εταιρική φύσης διαπραγμάτευση και ένα εταιρικού χαρακτήρα αποτέλεσμα. Εάν δούμε τι γίνεται με αυτές τις συμφωνίες στην Νότια Αφρική, εκεί μπορούμε να διαπιστώσουμε ξεκάθαρα ότι βεβαίως υπάρχουν κάποια ιστορικά προβλήματα όσον αφορά την Τελωνιακή Ένωση, αλλά από την άλλη υπάρχουν πολύ ξεκάθαρα ε, προβλήματα σε σχέση με τον τρόπο που κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή της διαπραγματεύσεις σε σχέση με την Νότια Αφρική. Γι' αυτό ε, πραγματικά αρνούμε να επιβάλλω αυτές τις ε, σχέσεις, τις εταιρικέ σχέσεις μέσα αυτή τη πίεση. Γιατί οι προθέσει αρχικά ήταν εντελώ διαφορετικέ. Θεωρώ ότι είναι έντιμο εκ μέρου του Ντέιβιτ να δώσουμε μία προθεσμία δύο ετών. Αλλά λόγω του ΠΟΕ δεν είναι δυνατόν να υπάρξει μια επαόριστον παράταση. Επιτρέψατε μου να συμμετάσχω σε αυτή τη συζήτηση, γιατί εγώ ηγούμαι τι ε, αντιπροσωπείε, με επικεφαλή αντιπροσωπεία για την Κένια και τη Ζάμπια. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι η παρούσα κατάσταση δεν μπορεί να εξακολουθήσει όχι επειδή είναι σύμβατη ήδη από το 2007, αλλά επειδή δεν είναι δίκαιοι απέναντι σε χώρες ε, που βρίσκονται στην ίδια κατάσταση αλλά που δεν επωφελούνται από το γενικευμένο σύστημα προτιμήσεων γιατί δεν ε, ανήκουν στις χώρες ΑΚΕ. Για παράδειγμα, οι χώρες της Λατινικής Αμερικής, στη γειτονία της ε, Ασίας που έχουν αντίστοιχες, ε, μια αντίστοιχη ανάπτυξη, παρόλα αυτά δεν μπορούν να αποφοληθούν από αυτό το εξαιρετικά ε, γενναιόδωρο σύστημα προτιμήσεων. Άρα πρόκειται για ένα ζήτημα εντιμότητος εκ μέρους ημών των Ευρωπαίων έναντι χωρών που θέλουμε να τις αντιμετωπίζουμε ισότιμα. Και αυτό είναι το ζητούμενο. Γι' αυτό πιστεύω ότι κατά την άποψή μου θα πρέπει να θέσουμε ένα τέλος στην παρούσα κατάσταση, είτε σε ένα χρόνο, είτε σε δύο χρόνια. Αυτό το αφήνω στην διακριτική ευχέρεια αυτής της Επιτροπής, αλλά θα υποστηρίξω σαφώς την πρόταση της Επιτροπής όσον αφορά το βασικό της στόχο, να πει ξεκάθαρα δηλαδή ότι αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί, θα πρέπει να πάυσει. Τώρα, ας ακούσουμε την Επιτροπή. Σάντρα Γκαλίνα, καλησπέρα. Θα επικεντρωθώ τροπολογία 1 και τροπολογία 3 στην παρέμβασή μου. Και στόχος μου είναι να είμαι σύντομη. Πρώτα απ' όλα σας ευχαριστούμε και για την έκθεση και για την ενδιαφέρουσα συζήτηση που δείχνει το ενδιαφέρον σας και είναι ενθαρρυντικό ε, για οποιονδήποτε εργάζεται πάνω σε ένα θέμα να βλέπει ότι υπάρχει ενδιαφέρον από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Λοιπόν, για την τροπολογία 1, Με όλο το σεβασμό διαφωνούμε, διότι έρχεται αυτή η τροπολογία σε αντίθεση με τις ιδεολογικές σκέψεις για την κατεξουσιοδότηση πράξης και επίσης είναι και διαφορετικό αυτό προτείνεται από τις τροπολογίες που είχαν προταθεί στο πλαίσιο Omnibus. Ίσως θα μπορούσα ακόμη να προσθέσω ότι οι σχέσεις μεταξύ Ευρωκοινοβουλίου και Κομισιόν για τις κατεξοσιοδότηση πράξη διέπονται και από τη συμφωνία πλαίσιο και από την κοινή συνεννόηση ή κατανόηση και γι' αυτό δεν θεωρούμε ότι θα πρέπει ad hoc να υπάρχουν συμπληρώματα σε αυτές τις ε, νομοθετικές πράξεις. Ε, τροπολογία επειδή είμαι λίγο σπασίκλα θα έλεγα στη λεπτομέρεια, για τα λουλούδια 7% το πολύ είναι και σε κορα όχι 23% το μέγιστο ποσοστό δασμών που του επιβάλλεται όταν μπαίνουν στην Ένωση για την ποτσόνα την Αμίμπια, την Νότια Αφρική είναι σαφέ ότι εκεί ε, υπάρχει κάποια προσωρινή εφαρμογή, κάποιο που ίσως να μην είναι και νομικός σταθερό. Η Νότια Αφρική όμως μέχρι ότου την DCA καλύπτεται πλήρως. Ε, υπάρχουν νομικέ ε, διατάξει. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε πολύ προσεκτικοί με το ποιο είναι ποιο, όπω και ο κύριο Φιέλνερ, ίσως να μην είναι το πρόβλημα απαραίτητα η Ναμίμπε, Μποτσουάν, Ευρωπαϊκή Ένωση, ίσω κάποιο άλλος να ευθύνεται. Για το πολύ καλό ερώτημα του κυρίου Ρινάλτη που λέει μπορούμε να προστατεύσουμε τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, ή και ακόμα πιο συγκεκριμένα τα συμφέροντα των χωρών ΑΚΕ. Ήμουν 12 χρόνια στη Γενέβη, άρα δεν υπάρχει παρέτηση δικαιώματος εκεί, δεν υπάρχει waiver. Για την Ταϊτή τώρα. Μπορούμε να αρχίσουμε συζητήσεις σε σχέση με τη δικαιοσύνη. Τι είναι δίκαιο, τι δεν είναι. Ότι ο νόμος διαφορές δεν αναγνωρίζει, ούτε χρώμα μαλλιών βλέπει, ούτε χρώμα ματιών. Άρα η IT ήταν ακριβώς στην ίδια κατάσταση, δεν υπήρξε κάποια διάκριση. Δεν μπορώ όμως ε, να το ε, ξεπετάξω το θέμα, αλλά είναι μια λιγότερα αναπτυσσόμενες χώρες, η ε, δεν είναι η μόνη όμως, υπάρχουν και άλλες ε, χώρες σαν την στις, μεταξύ των λιγότερων αναπτυγμένων χωρών και τι γίνεται και με αυτές. Λοιπόν, τροπολογία 3 και σας παρακαλώ να δείτε και την αιτιολογική έκθεση η οποία είναι προσαρτημένη στο ε, σχέδιο έκθεση, είναι πολύ καλογραμμένη και περιγράφει πολύ καλά το Μάρα σαν μια γεφυρωτική λύση, θα έλεγα. Πρέπει να αλλάξουμε τον αριθμό των χωρών που δεν έχουν ακόμη επικαιρώσει. Είναι 17 και όχι 18 πλέον και ελπίζουμε και έχουμε αισιοδοξία ότι τα επόμενα δύο χρόνια θα μειωθεί ακόμη περισσότερο αυτός ο αριθμός και θα μηδενιστεί. Στην, στο αιτιολογικό υπόμνη, λοιπόν, στην αιτιολογική έκθεση, είδα τη λέξη πίεση να επαναλαμβάνεται αρκετέ φορέ. Θα έλεγα ότι αυτό το οποίο έχουμε αυτή τη στιγμή μπροστά μας είναι μία όθηση. Μην μπερδεύουμε τα πράγματα. Θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο να πείσω τον Επιτροπό μου να πει ότι ορίστε έχουμε τώρα μία πρόταση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για να αλλάξει ένα νομοθέτημα μόνο και μόνο για να ασκήσουμε πιέσει στι διαπραγματεύσει. Αυτό δεν είναι απαραίτητα ορθό και σωστό, διότι η συλλογιστική που διέπει αυτή την νομοθεσία είναι η σχέση να ε, τοποθετηθεί σε ένα σωστό και σταθερό νομικό, αλλά και προβλέψουμε, θα έλεγα, νομικό πλαίσιο με όλε τι επιπτώσει που αυτό μπορεί να έχει. Στην επόμενη παράγραφο λέγεται η επιβολή μια τόσο σύντομη μονομερού προθεσμία. Κοιτάξτε, μπορούμε να το συζητήσουμε και είναι ενδιαφέρον να συζητούμε γιατί έχουμε ανταλλαγή απόψεων και στις ανταλλαγές απόψεων κανείς μπορεί να καταλήξει σε μια ορθή επιλογή, αν υπάρχει βέβαια ορθή επιλογή, όπως έλεγε και ο κύριος Ρινάλντι. Ξέρετε κάτι, δεν υπάρχει καν προθεσμία. Η προθεσμία έχει εκπνεύσει, ήταν το 2007. Α δούμε τις ε, συμφωνίες οικονομικές εταιρικές σχέσεις. Ε, την συμφωνία την είχαμε το 99 με τι χώρε ΑΚΕ, που το ζήτησαν. Είπαν 40 χρόνια σχέσεις όπου απλά εσείς μα δίνατε μονομέρειε που όχι. Εμεί θέλουμε τη δική μας ε, πραγματική εταιρική σχέση. Το 2000 έχουμε τη Συμφωνία Κοτονού. Και η αλληλουχία είναι πολύ ενδιαφέρουσα, γιατί όλοι εστιάζουν στον ΠΟΕ. Αλλά με επιτρέπετε να πω, δεν είναι η σωστή οπτική. Αυτό που διάλεξαν ε, ήταν το 1999 και όχι το 2000, χωρίς ιδιαίτερη πίεση, να επιλεγεί μια διαφορετική εταιρική σχέση. Έχουμε λοιπόν το κοτόνο το 2000, ήμουν παρούσα και στην Τόχα, όταν είχαμε αυτά τα περίφημα waiver και για τις μπανάνες, είχαμε τις διαπραγματεύσεις τότε, άρα τα ξέρω καλά. Και αυτή η προθεσμία το 2007 ήταν κάτι που πετύχαμε χάρη και στην πίεση των συναδέλφων της χώρας ΑΚΕ και ξέρετε προσπαθήσαμε, παλέψαμε για το 2007. την Κωνσταντίνα, από τις Φιλιππίνες, κάτι, κάτι βγάλαμε τέλος πάντων. Θα μπορούσα να σας πω και ονόματα ανθρώπων με σάρκα και οστά που μπορείτε να συμβουλευτείτε και έχουν μια άποψη για το 2007. Ίσως πράγματι υπάρχει ένα επίπεδο αλληλεγγύης μεταξύ των αναπτυσσόμενων χώρων. Αυτό δεν το αρνούμε. Αλλά ότι το 2007 δεν σημαίνει τίποτα για αυτούς που δεν είναι στον κόσμο, ε, που δεν ανήκουν στις περιοχές ΑΚΕ, νομίζω ότι δεν αληθεύει. Φτάνασαμε το 2008, εγώ τότε ήμουν στην Γενέβη και το είχα νιώσει. Τότε κάπως ε, ε περισπάστηκε η προσοχή μας γιατί υπήρχαν άλλα πράγματα, αλλά ήδη κάποιοι άρχισαν να μας κοιτάζουν το 2008 και οι εταίροι μας. Σας αφήνω λοιπόν να σκεφτείτε, έχοντας μπροστά μας τον ορίζοντα του 2014, ο Επίτροπος μου πώς θα κάνει αυτό το άλμα και πώς θα πει, ναι, δίνομαι χρόνο για να γίνουν κάποια πράγματα. Και να σας πω κάτι, αν θέλαμε έστω και για ένα χρόνο να το αναβάλουμε. Εγώ δεν είναι... Ε, δεν το λέω για ως αστείο. Δεν έχουμε τελικά μία πολιτική συνοχή. Γιατί ξέρετε και από το ποια χώρα έχουμε μπροστά μας. Γιατί είναι διαφορετική η μεταχείριση. Έχουμε την τάδε χώρα, της δίνουμε μία συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης, ακόμα και αν δεν είναι χώρα ε, με ελάχιστα αναπτυγμένη. Υπάρχει ασυμμετρία, κάτι πολύ χρήσιμο για τις χώρες ΑΚΕ, αλλά αυτό το αποφθαλμιούσαν και κάποιοι από τους εταίρους μας ε, στην Κεντρική Αμερική που δεν το πέτυχαν. Ούτε τη συσσόρευση την πέτυχαν που είναι μια λιμουζίνα αν θέλετε ή ένα πολύτιμο παιχνίδι που συνοδεύεται όμως μόνο από τις συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης. Άρα έχουμε δύο παραμέτρους, κάλυψη προϊόντων και όροι, προποθέσεις που άλλαξαν. Και υπήρχε διαφορετική μεταχείριση των ε, χωρών ΑΚΕ. Και δεν υπήρξε ποτέ εκ των προτέρων εφαρμογή πριν υπάρξει επικύρωση. Ναι, μπορείτε να συντομεύετε παρακαλώ. Ναι, μάλιστα. Θέλω να εστιάσω και σε κάτι άλλο. Στην ουσία ουσιαστικά των διαπραγματεύσεων. Στην αιτιολογική έκθεση διαβάζω εάν επιληθούν όχι αυτά τα ζητήματα. Δεν νομίζω ότι είναι προ το συμφέρον τη Ευρωπαϊκής Ένωσης να ολοκληρώνει συμφωνίες που δεν ικανοποιούν τους ε, συμβαλωμένου. Ούτε έχει γίνει, ούτε θα γίνει κάτι τέτοιο. Άρα τελικά αυτά τα δύο χρόνια είναι χρήσιμα. Δεν είναι όμω και κατά ανάγκη απαραίτητα. με αναβολή κατά ένα χρόνο, τι κάνετε ουσιαστικά. Πονομεύετε την όθηση που έχει ήδη δημιουργηθεί. Γιατί δεν μιλάμε για πιέσεις, μιλάμε για όθηση, μιλάμε για μία, ένα αριθμό που έχει πάρει το πράγμα. Και πιστεύω ότι υπάρχει οριμότητα σε όλα τα κράτη. Νομίζω ότι θα πρέπει λοιπόν να ενισχύσουμε και όχι να υπονομεύσουμε με πιέσεις. πρέπει να δείτε και την κατάσταση στο εσωτερικό των ε, εταίρων μας από τις χώρες ΑΚΕ και ιδίως στην Αφρική. Επίσης, ετέθε ένα ζήτημα για, το, για την εντιμότητα και τη δικαιοσύνη. Ποιοι υπέγραψαν, έκαναν την προσπάθεια και ποιοι δεν έκαναν την προσπάθεια. Εγώ θα σας πω μια ιστορία. Σύντομη ιστορία, παρακαλώ. Ναι, για δύο χώρες όμως που είναι στον, στην ίδια περιοχή ΑΚΕ. Μία χώρα δεν επέλεξε το 2007 την ΕΠΑ, γιατί είπε πολύ ειλικρινά ότι δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να αντιμετωπίσω τις δεσμεύσεις αυτές. Η άλλη χώρα, δίπλα, προχώρησε. Υπέγραψε. Απλά. Δεν έχει ακόμη επικυρώσει. Κρεμεί. Οι δύο χώρες αυτές, την 1η Ιανουαρίου του 2014, αν παραταθεί βέβαια προθεσμία, θα είναι σε μια κατάσταση, μιλάω για την Καμπόν και το Καμερούν. Το Καμερούν θα έχει άλλο ένα χρόνο τις προτιμήσεις χωρίς να έχει κάνει τίποτα, απολύτως τίποτα διαφορετικό από την Καμπόν, παρά το ότι απλά υπέγραψε μια συμφωνία, ενώ η Καμπον το 2007 δεν προχώρησε με συμφωνία οικονομική εταιρική σχέση, σήμερα πληρώνει δασμούς και θα πληρώνει με φεν ε, δασμούς το 2014. Γιατί το GSP θα αρχίσει να ισχύει από την 1η Ιανουαρίου του 2014 κατά πάσα πιθανότητα. Με αυτή την πολύ σύντομη ιστορία λοιπόν βλέπετε πολύ καλά ότι οι δράσεις μας ως Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι ουδέτερε, Ακόμη και ένα επιπλέον έτος θα δημιουργήσει πολύ ε, σοβαρέ από πολιτική πλευράς ε, ανισότητες. Δημιουργούνται λοιπόν αθέμητο ανταγωνισμός ε, και άλλα προβλήματα. Τελικέ παρατηρήσει του εισηγητή David Martin. Ο Keith Taylor είπε ότι είχε την εντύπωση πώ δεν ήμουν αντίθετο σε μια άνευ καταληκτηρίου ημερομηνία ε, συνέχιση ισχύω αυτού του κανονισμού. Και θα πρέπει να πω, αφού άκουσα την απόψηνή συζήτηση, πω ίσω να μην κάνει λάθο, γιατί Ακούσαμε μόλις από την Κομισιόν που ξεκίνησε ότι ναι, τώρα είναι η ώρα, αλλά τελικά κατέστησε σαφές ότι πρόκειται για άσκηση πίσης προς τις χώρες ΑΚΕ για να υπογράψουν μια συμφωνία για την οποία μπορεί να μην είναι έτοιμοι να την ε, ε, συνυπογράψουν. Αν πιστεύουμε λοιπόν σε όλα αυτά και θα πρέπει να σας πω ότι τυχαίνει, την χάνει να το πιστεύω γιατί ήμουν εισηγητής για δύο από τις επιτυχείς ε, συμφωνίες για την Καρεβική και τον Ειρηνικό. Μπορούμε να πούμε ότι είναι άδικο για τις χώρες που υπέγραψαν τις ε, συμφωνίες. Ε, αυτές τις υπέγραψαν γιατί υποτίθεται είναι καλό για αυτές. Αν όμως ε, τελικά τις υπέγραψαν γιατί τους ασκήθηκε πίεση, τότε αλλάζει η υπόθεση. δεν μιλάω για δικαιοσύνη για για τους όσους υπέγραψαν τις συμφωνίες. θεωρώ πως αυτοί που τις υπέγραψαν, τις υπέγραψαν διότι πιστεύουν ότι είναι προς το συμφέρον της, του οικονομικού συμφέροντος της χώρας τους πιο στεναρό, πιο ισχυρό επιχείρημα είναι η συμβατότητα με τον ΠΟΕ και γι' αυτό και τελικά μίλησα για τελική εκπνοή. Αλλά τι είναι το μαγικο πρωτη Πρώτου 2014, γιατί τι διαφορά κάνει από την πρωτη η Πρώτου 2013 ή 12 και γιατί να μην γίνει το 2016. Αυτό που κάνει η Κομισιόν δεν έχει περισσότερο νόημα από οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία, εκτός φυσικά από την άσκηση πίεσης στις χώρες ΑΚΕ στις, που έχουν ή δεν έχουν υπογράψει τις συμφωνίες τους. Εγώ δεν θα ήθελα αφρικανικές χώρες να υπογράψουν ε, για συμφωνίες με τις οποίες δεν είναι άνετοι. Θέλω καλύτερα να έχουν χρόνο να διαπραγματευτούν. Εάν μέχρι το τέλος του 2016 δεν μπορούν να καταφέρουν να το κάνουν αυτό, τότε θα πρέπει να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες εναλλακτικών οικονομικών καθεστώτων. Πάντως δεν θα πρέπει να επιμείνουμε ώστε να ολοκληρώσουν τις διαπραγματεύσεις. Όταν θα περάσει αυτό εδώ, θα ξέρουν ακριβώς πόσους μήνες θα έχουν διάθεσή τους για να διαπραγματευτούν ακόμη. Αυτό θα τους δώσει κάτω από ένα χρόνο, γιατί ο κανονισμός αυτός ούτως ή άλλως ε, ε γύρω στο φθινόπωρο θα εγκριθεί οριστικά αν εγκριθεί. Να πω κάτι ακόμα. Όχι για να γκρινιάξω, αλλά για να πω ε, για το πρόβλημα του ότι δεν ενημερωνόμαστε επαρκώ για την, για την, ε, για την ε, συμφωνία. Ξέρω πω η Μποτζοάνα πρόσφατα υπέγραψε συμφωνία, η Ζιμπάμπουε, συγγνώμη. Δεν ενημερώθηκα όμω από την Κομισιόν. Εγώ λέω 18 18 χώρε δεν έχουν υπογράψει. Ε, αυτή είναι η θέση μα στο Κοινοβούλιο, αυτό ξέρουμε. Επισήμω δεν ήρθε κανεί να μα ενημερώσει, να μας πει ότι η Ζιμπάμπο υπέγραψε την συμφωνία. Όντω έτσι είναι. Σας ευχαριστώ για τη συζήτηση. Η ημερομηνία για την υποβολή είναι 18 Μαΐου, η υιοθέτηση στην Επιτροπή 18 Ιουνίου και προσθενότατα στην Ολομέλεια θα περάσει από το Σεπτέμβριο το θέμα. Σημείο 23. Αντιπροσωπεία στην Ανατολική Αφρική. Η επίσκεψη αυτή ήδη αναφέρθηκε. Έχετε την σχετική έκθεση στους φακέλους σας. Το μόνο πράγμα που θα μπορούσα να πω, συνοψίζοντας, είναι ότι ήταν πολύ ε, αυτή η επίσκεψη. Σχόλια. Ε, item 24. Officially support. Σημείο 24. εφαρμογή του κανονισμού για τις εξαγωγικές πιστώσεις που την χάνουν δημόσιας στήριξης. Εισηγητή μα ο Γενίκη Ζανό, που ήταν και εισηγητή για το νομοθετικό φάκελο και θα του δώσω αμέσω τον λόγο. Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω πω είναι ένα καλό νέο που κάνουμε αυτή τη συζήτηση, γιατί όντω αφού το Κοινοβούλιο έχει την συναπόφαση για την εμπόριο, είναι σημαντικό να παρακολουθούμε την εφαρμογή των ε, κανονισμών οδηγιών που διαπραγματευόμαθα και που υιοθετούνται. Θα ήθελα να εκφράσω την χαρά μου γιατί είναι στην αίθουσα εκπρόσωποι της Κομισιόν και έπειτα εκπρόσωποι της Γραμματείας του Συμβουλίου Ιδιαίτερα αυτοί οι οποίοι συμμετέχουν στην ομάδα διαπραγματεύσεων για τις πιστώσεις εξαγωγών και που θα μπορέσουν, ελπίζω, να συμμετέχουν στην ανταλλαγή απόψεων. Βέβαια, η συζήτηση αυτή είναι πολύ συγκεκριμένη γιατί η εφαρμογή αυτού του κανονισμού οδηγεί στο ότι τα κράτη-μέλη τώρα πρέπει να έρθουν με ένα έγγραφο Ε, που θα αναφέρει τα όσα έχουμε συμφωνήσει και είναι ενδιαφέρον να συζητήσουμε για τα πράγματα αυτά μέσα στο πλαίσιο του Συμβουλίου. Ε, να δούμε τι συμβαίνει εκεί. Είναι σημαντικό, αν θυμάστε και τη συζήτηση που κάναμε, Είναι σημαντικό η Κομισιόν στις σχέσεις με τους ε, εμπορικούς μας εταίρους ε, να φέρει αυτό το, το διακύβημα του ισότιμου πεδίου όσον αφορά τις υπηρεσίες ε, τους φορείς εξαγωγών και αναβάλαμε τη συζήτηση γιατί πριν από λίγες εβδομάδες η, Κομισιόν ήταν στην Κίνα για να συζητήσουν για ένα μνημόνιο συμφωνίας με την Κίνα και με το ΕΣΥΠΑ εκτός του ΩΣΑ ακριβώς από αυτού του θέματος. Και έπειτα θα θυμάστε, Πρόεδρε, έχετε στις 3 ε, Ιανουαρίου στείλει μια επιστολή στο όνομα αυτής της Επιτροπής στην Προεδρία, τη Δανική, ακριβώς γιατί διαπιστώναμε ήδη τις δυσκολίες εφαρμογής των όσων είχαμε διαπραγματευτεί και υιοθετήσει. Ποιο είναι λοιπόν το σημείο που δημιουργεί πρόβλημα. Αυτό που δημιουργεί πρόβλημα στο πλαίσιο του Συμβουλίου και θα είναι ενδιαφέρον να ακούσουμε τα σχόλια είναι ακριβώς αυτή η ιδέα ότι οι φορείς των ε, πιστώσεων εξαγωγών είναι μέρη της ε, επιτροπής μας Έχουμε υιοθετήσει συμφωνία, έχουμε υιοθετήσει συμφωνία με την Ουγγρική Προεδρία ε, που λέει ότι οι δραστηριότητε των ε, φορέων ε, πιστώσεων εξαγωγής θα πρέπει να συμμορφώνονται προς τις γενικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα θέματα εξωτερικής δράσης, δημοκρατία, ανθρώπινα δικαιώματα, συνοχή για την ανάπτυξη. Έμεσα λοιπόν λέγαμε ότι ε, το τμήμα των, της αναφοράς, το reporting, θα πρέπει να συμμορφώνεται προς το άρθρο 21 της συνθήκης. Δυστυχώς, όταν βλέπουμε το πρώτο σχέδιο, που μπορέσαμε να έχουμε από τους Βρετανούς και σας, δεν σας λέω τις λεπτομέρειες, το βλέπετε και από μακριά, είμαστε σε ένα είδος, αφήστε τις ε, βρετανικές ε, ε, πτυχές, αλλά για τις πτυχές έκθεση που εμείς θεωρούμε σημαντικές είμαστε σε ένα είδος κενού, απόλυτου κενού, που μας ανησυχεί βεβαίως, γιατί... Το Κοινοβούλιο για μια ακόμα φορά είναι σε διαπραγμάτευση με την Προεδρία, με το Συμβούλιο και θεωρήσαμε πως ήταν σημαντικό. Από τη στιγμή που οι υπηρεσίες εξωτερικών πιστώσεων ε, εμπίπτουν ε, στην ε, δημόσια σφαίρα, δηλαδή είναι δημόσιο χρήμα, θα έπρεπε να συμμορφώνονται και στους στόχους Τη Ένωση. Ε, είναι καλό λοιπόν που γίνεται αυτή η συζήτηση σήμερα, ώστε να γνωρίζουμε τώρα σε αυτή τη φάση κλειδί όπου τα κράτη-μέλη πρέπει να δώσουν τι πρώτε εκθέσει, όπου γνωρίζουμε ότι θα χρειαστουν δυο δύο-τρία χρόνια για να επιτύχουμε τα αποτελέσματα που υπολογίζαμε στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, αλλά να εξασφαλίσουμε ότι τουλάχιστον το πρώτο χρόνο θα υπάρχει βούληση ακόμη μια φορά στην άσκηση του reporting να συμμορφωθούν στην συνθήκη της Ένωσης και στους στόχους της Ένωση. Σας ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ. Δεν χρειάζεται να υπογραμμίσουμε ακόμη μια φορά την σημασία αυτή της προσπάθειας. Να πάμε άμεσα στην Κομισιόν. Πάολο Γκαρζώτη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η εξολόγηση του εισηγητού είναι αρνητική, έτσι δεν είναι. Ναι, αλλά τον ευχαριστώ παρόλα αυτά, γιατί είναι επικοδομητική πάντοτε. Δεν είναι μια αξιολόγηση, γιατί δεν έχουμε ακόμα στα χέρια μας την έκθεση. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή όχι μόνο για την εργασία που έκανε όσον αφορά την έγκριση της πρότασης, αλλά για την επικοδομητική του άποψη όσον αφορά το πότε θα πρέπει να συνταχθεί η έκθεση αυτή. Συμφωνήσαμε για το χρονοδιάγραμμα. Τον Ιούλιο οι χώρες μέλη θα πρέπει να δώσουν την πρώτη του ετήσια έκθεση για το 2011 και στη συνέχεια η Επιτροπή θα πρέπει να κάνει μια αιτήσια επιθεώρηση του Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στη βάση το, αυτών των πληροφοριών καθώς και μια αξιολόγηση ε, εν σχέση με τους ε, φορείς των πιστώσεων εξαγωγών. Και η Επιτροπή θα προσπαθήσει να εξασφαλίσει ότι εφαρμόζεται σωστά ευρωπαϊκή νομοθεσία και θα κάνουμε μια σχετική αναφορά, έτσι όπως προβλέπετε. Τώρα, όσον αφορά το περιεχόμενο, δηλαδή το πώς θα πρέπει να κάνουν αυτή την αναφορά οι χώρες μέλη και πώς θα πρέπει να κάνει την αναφορά αυτή η Επιτροπή, είπα ότι το πρώτο τμήμα του παρατήρηματος 1 λέει ξεκάθαρα τι θα πρέπει να αναφέρουν οι χώρες μέλη σύμφωνα με το εθνικό τους ε, πλαίσιο όσο αφορά τις ευθύνες κλπ. Ε, το Συμβούλιο θα πρέπει να παράσει ένα κατάλογο εργαλείων για να διευκολύνει το έργο αυτό, ούτε ώστε να εξασφαλίσουμε ότι έχουμε την αναγκαία τις αναγκαίες πληροφορίες, αναγκαία δεδομένα για να κάνουμε αυτή την ετήσια επισκόπηση και αυτός ο κατάλογος θα συζητηθεί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με τον εισηγητή και πιστεύουμε ότι θα είμαστε σε θέση στη βάση μιας καλής βούλησης των χωρών μελών να έχουμε μια ετήσια επιθεώρηση η οποία θα είναι αρκετά ικανοποιητική για το Κοινοβούλιο και, και θα προβούμε σε μια αξιολόγηση της ε, συμμόρφωσης. Εάν δεν έχουμε όμως αρκετά δεδομένα για να γίνει αυτή η αξιολόγηση, απλούστατα θα πρέπει να λάβουμε γνώση αυτής της έλλειψης. Αλλά από αυτά που διαπιστώσαμε σήμερα στη συζήτηση που έγινε στο Συμβούλιο, έχω, έχω την πεποίθηση ότι θα είναι επαρκή οι πληροφορίες, τα δεδομένα ε, ίσως όχι την πρώτη φορά όπως είπε ο συγκητής, γιατί αυτό δεν είναι εύκολο, γιατί πρόκειται για ένα καινούριο πεδίο για όλους μας, αλλά είμαι σίγουρος ότι θα είμαστε σε θέση να καταλήξουμε σε μια αμοιβαία συνεννόηση. Και θα ήθελα να καταλήξω λέγοντας ότι είναι ακόμα νωρίς, δεν έχουμε ακόμα τις εκθέσεις. Ίσως ε, αργότερα γύρω στο τέλος του χρόνου θα μπορούμε να έχουμε μια άλλη συζήτηση. Ο εισηγητής είπε επίσης πόσο σημαντικές οι νέες εξελίξεις ε, στον τομέα των πιστώσεων εξαγωγών ε, ε, μεταξύ Κίνας και είπα όταν ο πρόεδρος της Κίνας επισκέφθηκε τον πρόεδρο Ομπάμα συμφώνησαν σε μια κοινή δήλωση ότι θα αναλάβουν πρωτοβουλία να διαπραγματευθούν τις ε, διεθνείς κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά τις πιστώσεις εξαγών και να καταλήξουν μια συμφωνία το 2014. Πήγαμε ήδη στην ε, Κίνα ε, και θεωρούμε ότι η Κίνα είναι ε, ιδιαίτερως ε, κάπως επιφυλακτική όσον αφορά αυτές τις συζητήσεις με τις Ηνωμένε Πολιτείες. Ελπίζουμε να μάθουμε περισσότερα πράγματα μετά τη συνάντηση που θα γίνει αρχές Μαΐου μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας, ούτως ώστε να μπορούμε να διευκρινίσουμε καλύτερα το χρονοδιάγραμμα αυτών των διαπραγματεύσεων, αλλά θα είναι πολύ σημαντικό από οικονομική πλευρά, γιατί θα είναι η πρώτη φορά που θα μπορέσουμε κατ' ουσία να συζητήσουμε τις πιστώσεις επί των εξαγωγών με τους ε, Κινέζους εταίρους μας και θέματα τα οποία βρίσκονται υποσχέτως σε αυτήν την έκθεση, το περιβάλλον, εργαστικές συνθήκες κλπ. Ε, θα είναι πολύ δεύτερα να συζητηθούν με την Κίνα και βεβαίω θα πρέπει να επιτευχθεί μια ισορροπία σε σχέση με τη σημασία και τον ουσιαστικό ρόλο αυτών των αρχών και καθώς και της οικονομικής ε, βαρύτητας που έχει η Κίνα στο τραπέζι της συζήτησης για τις πιστώσεις εξαγωγών. Κάτι όπως την ενδιαφέρον για την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόεδρος, έχω ένα αίτημα εκ μέρους του Συμβουλίου. Δεν ξέρω γιατί δεν θα έπρεπε να ακούσουμε το Συμβούλιο, τη Γραμματεία, του κύριο Ανδρέα Στρούμπ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε δεν ήταν έτοιμα, αλλά μου ζητήθηκε κατά πώς θα μπορούσα να δώσω κάποια ένδειξη εφόσον ο πρόεδρος της ομάδας για τις πιστώσεις εξαγών δεν μπορούσε να παραβρεθεί εδώ. Θα ήθελα απλώς να σε επικυρώσω ότι λάβαμε την επιστολή σας. Σε ευχαριστούμε πολύ. Αυτό το οποίο συμβαίνει είναι καινούριο και εμφανές για όλους μας και για τις χώρες μέλη. Και εγώ προσωπικά είμαι πιο αισιόδοξο από τον κύριο Ζαντό, εάν μου το επιτρέπετε. Αλλά όπως είπε ο συνάδελφος από την Επιτροπή θα πρέπει να αναμένουμε για να δούμε ποια θα είναι τα αποτελέσματα την ενταντιγμένη στιγμή. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα οι καταληκτήριες παρατηρήσεις από τον εισηγητή. Κ. Ζαντώ, ευχαριστώ πολύ τον εκπρόσωπο τους εκπρόσωπους της Επιτροπής και τον εκπρόσωπο του Συμβουλίου γιατί θεωρώ ότι είναι σημαντικό να μπορούμε να συζητήσουμε για την υλοποίηση αυτού που συζητούμε, διαπραγματευόμαστε σήμερα και να έχουμε μια εκ του παρακολούθηση των συμφωνιών που περνάμε. Γιατί ε, ακόμα και σε αυτή την Επιτροπή, πώς να το πω, βρισκόμαστε σε μια διαδικασία εκμάθησης της διαδικασίας συναπόφασης και είναι σημαντικό να βλέπουμε πώς γίνονται τα πράγματα στην πραγματική ζωή. Ευχαριστώ πολύ τους συναδέλφους από την Επιτροπή και το Συμβούλιο που ήρθαν. Ευχαριστούμε. Τελευταίο σημείο άκτα, το σημείο υπαριθμών 25. Όπως ξέρετε, πρόκειται για μια διεθνή συμφωνία, πολυμερή. Είμαστε η αρμόδια επιτροπή, ο συγητής μας είναι ο κύριος Ντέιβιτ Μάρτιν. Ε, είχαμε μια προηγούμενη ανταλλαγή απόψεων και τώρα έχουμε το στέγιο σύστασης ε, εκ μέρους του εισηγητού. Βρίσκεται στα έγγραφά σας. και ο εισηγητής ε, προτείνει, από το, προτείνει στο Κοινοβούλιο να μην δώσει τη συγκατάθεσή του σε αυτή τη συμφωνία. Πριν δώσουμε το λόγο στον εισηγητή, Επιτρέψατε μου να σας πω ε, ε, ε, λόγω του αιτήματος κάποιων επιτροπιών που γνωμοδοτούν και μας ζήτησαν να περιμένουμε τη δική τους γνωμοδότηση, αποφασίσαμε να κάνουμε μια αλλαγή στο χρονοδιάγραμμά μας και γι' αυτό η ψηφοφορία θα λάβει χώρα κατά τη διάρκεια της συνεδρίασής μας τον Ιούνιο και όχι το Μάιο. Έτσι, ούτως έχουν λοιπόν, ούτως έχει το χρονοδιάγραμμα. Η ψηφοφορία θα γίνει στην ίντε. Και τώρα θα περάσουμε στη συζήτηση του σχεδίου σύστασης ακούγοντας πρώτα τον εισηγητή μας, τον David Μάρτιν. Έχεις το λόγο, David. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Έχουμε εσείς το θέμα αυτό κατ' επανάληψη, άρα δεν χρειάζεται να επισέλθουμε σε πολλές λεπτομέρειες. Αλλά όπως είπες, μετά από πολλές διαβουλεύσεις, εγώ αποφάσα να συστήσω στην Επιτροπή να απορρίψουμε το άκτα. Και θα ήθελα να καταστήσω σαφές ότι δεν απορρίπτω την ανάγκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση να προστατεύσει την πνευματική της ιδιοκτησία και άλλωστε το είπα κατά επανάληψη σε αυτή την Επιτροπή ότι η Ευρώπη δεν είναι καλώς ε, εξοπλισμένη με πρώτε ύλε. Δεν μπορούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί στι πρώτε ύλε, αλλά θα πρέπει να είμαστε ανταγωνιστικοί όσον αφορά την καινοτομία και την δημιουργικότητα. Και αν θέλουμε να το κάνουμε, θα πρέπει να μπορούμε να προστατεύσουμε την πνευματική μα ιδιοκτησία σε μια παγκόσμια κοινωνία εγώ θεωρώ ότι δεν το επιτυχάνει, δεν επιτυχάνει αυτό το στόχο για άκτα. Γι' αυτό αποφάσισα να προτείνω να την απορρίψουμε, αλλά δεν ήταν μια εύκολη απόφαση. Ε, η άκτα θεωρώ ότι συγχαίει τα πάντα και θεωρώ ότι είναι σφάλμα στην ίδια συνθήκη να έχουμε ε, πνευματικά αγαθά και υλικά αγαθά. Και νομίζω ότι η Επιτροπή ε, συγχαίει τα πράγματα, τα θέτει εσφαλμένα. Ε, δεν είναι συγκρίσιμες αυτές οι δραστηριότητες. Η εμπορική παραποίηση και διαδικτυακή πειρατεία. Ε, είναι ελλειπής η ακρίβεια της άκτα για παράδειγμα όσον αφορά τις εμπορικές ε, ε, δεξιότητες. Δεν ξέρω τι σημαίνει κάτι τέτοιο, commercial skill, η κατάχρηση των εμπορικών δεξιοτήτων. Α, ε, της εμπορικής, συγγνώμη, της εμπορικής κλίμακας, συγγνώμη. Είναι αόριστος ο ορισμός της εμπορικής κλίμακας, commercial scale. και ε, ε, δεν ξέρω τι σημαίνει η εμπορική κλίμακα η οποία τελικά οδηγεί σε μια ποινικοποίηση. Η άλλη βασική ανησυχία είναι η υποχρέωση για τους παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών. Αλλά και εν πάση περιπτώσει ε, υποχρέωση μάλλον να προσφεύγουν ε, σε περίπτωση ε, παρανόμων, παραβίασης των δικαιωμάτων εκ μέρους παρανόμων παρόχων δεν νομίζω ότι θα πρέπει να επιβληθεί μια άμεση υποχρέωση στους ε, παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών να ε, πατάξουν την πειρατεία. Είναι δύσκολο να πείσει κανείς τους Κινέζους ή τους Ινδούς, για παράδειγμα, να υπογράψουν μια τετοια είδους συμφωνίας αλλά νομίζω ε, και νομίζω μια τέτοια συμφωνία ε, δεν πρόκειται να τους συγκεντρώσει τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Νομίζω ότι θα πρέπει να κοιθούμε μέσω World και άλλων οργανισμών. Ε, δεν ξέρω αν θα τα καταφέρουμε φέτος, του χρόνου ή σε μερικά χρόνια, αλλά τελικά θα τα καταφέρουμε και θα έχουμε μια συμφωνία η οποία θα είναι εφαρμόσιμη. και ε, δεν θα στρέφεται ε, εναντίον ορισμένων χωρών. Λοιπόν, όπως σας είπα, δεν ε, απορρίπτω την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας και ελπίζω ότι η Επιτροπή θα υποβάλει κάποιες προτάσεις για τη βελτίωση της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας όσον αφορά την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας αλλά δεν νομίζω ότι η συμφωνία αυτή είναι ο ενδεικμένο δρόμο. Η σκιώδης τώρα, πρώτος ο Κρίστοφερ από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον Ντέιβιντ για την παρουσίαση. Πρέπει να πω ότι με ένα μέρος της συζήτηση που γίνεται για την άκτα, έτσι δεν είμαι τόσο άνετος για αρκετούς λόγους κυρίως όμως γιατί η όλη συζήτηση έχει περιστραφεί μόνο γύρω από το θέμα ότι η άκτα είναι το πρόβλημα. Άρα την άκτα την πολεμάμε, την καταργούμε, αλλά αν κάποιο πάρει λίγη απόσταση θα καταλάβει ότι το πρόβλημα δεν είναι η άκτα αλλά η πειρατεία. Και το πρόβλημα είναι πώ θα, προστατεύσουμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα δικαιώματα πνευματική ιδιοκτησία. Το να επικεντρωνόμαστε μόνο σε αυτή την ε, συνθήκη βάζει την ουσία στο δεύτερο πλάνο. Και κατ' εμέ σημασία έχει πώ θα προστατεύσουμε τις θέσεις εργασία αν θα μπορέσουμε να προστατεύσουμε τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, αν θα καταπολεμήσουμε τα παραπημένα φάρμακα, τις απομιμήσεις ανταλλακτικών εξαρτημάτων κτλ. Δεν νομίζω ότι σκοτώνοντας, αν μου επιτραπεί έκφραση, την άκτα, κερδίζουμε τη μάχη. Όσοι έχουν παρακολουθήσει τι διαπραγματεύσει και τι συζητήσει, παραδείγματο χάρη για τη Συμφωνία Ελευθέρωση Συναλλαγών με την Ινδία, για παράδειγμα, και έχουμε και το διάλογο με την Κίνα. Ε, νομίζω ότι καταλαβαίνουν ε, ότι οι προσπάθειές μας να ε, τους κάνουμε να δείξουν μεγαλύτερο σεβασμό για τα πνευματικά δικαιώματα και να υιοθετήσουν πιο αυστηρή νομοθεσία. Δεν θα γίνουν πιο εύκολες οι προσπάθειές μας λοιπόν εάν εμείς έχουμε μια τέτοια ε, σύμφωνια που βασίζεται στο κοινοτικό και στο κεκτημένο μάλλον και μετά λέμε όχι δεν το θέλουμε αυτό. δεν θα βοηθήσει το να σκοτώσουμε την άκτα, το να τη θάψουμε αυτή τη συμφωνία. Ε, ακούω και διάφορες εναλλακτικέ. Όταν μπορούσαμε να είχαμε κάνει το ένα, θα μπορούσαμε να κάνει το άλλο. Και πραγματικά είναι ένας ειλικρινής ε, τρόπος να δει κανείς τι εναλλακτικέ υπάρχουν. Αν όμως ε, σκάψουμε κάτω από την επιφάνεια, θα δούμε ότι δεν πρόκειται για πραγματικέ εναλλακτικέ. Αν πούμε ότι πρέπει να πάμε πολυμερό, να το κάνουμε μέσω του ΠΟΕ. Νομίζω ότι το έχουμε προσπαθήσει λίγο πολύ. Αλλά δεν έχω ακούσει καμία σοβαρή πρόταση και ούτε και οι σοσιαλιστέ ήδη νομίζουν ότι μια συμφωνία με την Ινδία και την Κίνα στο πλαίσιο του ΠΟΕ, παραδείγματο χάρη, θα έδινε κάποια αποτελέσματα ω προ αυτή την πτυχή. Και κάποιοι λένε πρέπει να είναι πολυμερής γιατί δεν καλύπτει όλη την Ήπειρο. Ξέρετε, καλύπτει όμως το 50% του παγκόσμιου εμπορίου. Και αν το πρωτόκολλο του Κιώτο κάλυπτε το 50% των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα, θα ήμουν πολύ πιο χαρούμενος από το σημερινό ποσοστό του 26% που δεν περιλαμβάνει τις χώρες που κυρίως κάνουν αυτή την ε, πειρατεία. Το πρωτόκολλο του Κιώτο όμως δεν το θάψαμε, Κάποιους δεν αρέσει σε κάποιους το κεκτημένο, κάποιοι θέλουν μια τελείως διαφορετική προσέγγιση. Θα μπορούσαμε όμως να κάνουμε μια σύγκριση και πάλι με την κλιματική αλλαγή και το πρωτόκολλο του Κιώτο. Δηλαδή κάποιοι που ε, θα διαφωνούσαν πάρα πολύ με το πρωτόκολλο του Κιώτο. Εγώ νομίζω ότι υπάρχει ένα σημείο συνάντησης. Έχουμε ακούσει πολλά από τους ίδιους βέβαια κυρίως ανθρώπους. Σας πάντων ακούγονται διάφορες φήμες και κάποια πράγματα δεν μπορούν να τεκμηριωθούν από όσα ακούγονται. Έχω διαβάσει πολύ προσεκτικά, έχω ακούσει πάρα πολύ προσεκτικά και τι να σας πω, και η γλώσσα είναι ασαφής. Θα έπρεπε να είναι πιο ξεκάθαρο τι σημαίνει και τι επιπτώσεις θα έχει. Και σίγουρα και εγώ έχω θέματα με την άκτα. Όταν το μελετήσαμε το θέμα στο πλαίσιο του ΕΛΚΑ υπήρχαν τουλάχιστον δύο ξεκάθαρα σημεία που τα αφήξατε κι εσείς και τα οποία χρήζουν προσοχής. Το πρώτο είναι αυτή η έννοια commercial scale, εμπορική κλίμακα. Πώς ορίζεται και τι συνέπειε ε, υπάρχουν. Το ίδιο ισχύει με το άρθρο νομίζω είναι το 27 για τις συνθήκες υπό τις πίεση, οι πάροχοι ISPs πρέπει να δίνουν πληροφορίες για άτομα που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες τους και παραβιάζουν τα πνευματικά δικαιώματα, τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Είναι σαν να ζητάμε από έναν εξωγήινο να ζητάει από ένα γήινο δικαστήριο να επιληφθεί. Δεν είναι ξεκάθαρο για μένα αυτό. Πρέπει να έχουμε κατά νου ότι το να θάψουμε την άκτα δεν θα μας βοηθήσει. Καλύτερα θα τα προσπαθήσουμε να φτιάξουμε ε, τη συμφωνία αυτή. Μα κάποιος μπορεί να σας πει, κάποιος νοήμων θα σας πει, το κοινοβούλιο δεν μπορεί να κάνει τίποτα πέραν του να πει να ναι ή να όχι. Δεν μπορεί ούτε να τροποποιήσει την πρώτη, ώστε να προτείνει ένα κανονισμό, ο οποίο θα θεσπίζει τις διατάξεις και τα λοιπά ή θα ορίζει την εμπορική κλίμακα, για παράδειγμα. Αυτό πρέπει να είναι σαφέ. Εμεί δεν έχουμε τέτοια αρμοδιότητα. Δεν μπορούμε να το κάνουμε. Άρα το πιο ειλικρινέ και έντιμο που μπορούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι να στείλουμε πίσω τον μπαλάκι στου διαπραγματευτέ αυτή τη συμφωνία. Αυτοί που μα έδωσαν το κείμενο πρέπει να ξέρουν ότι δεν μα ικανοποιεί το χύψη ωμέγα μετά μπορεί να μα πούν βέβαια δεν μπορούμε να επαναδιαπραγματευτούμε, δεν μπορούμε να διορθώσουμε κτλ. Το έχω ξανακούσει βέβαια αυτό παραμύθι. Πάρα πολλέ φορέ ε, στο κοινοβούλιο μου παρουσίασαν ένα έγγραφο και μου είπαν πε ναι ή όχι, δεν μπορεί να αλλάξει τίποτα στο έγγραφο. Δεν τα πιστεύω αυτά τα πράγματα. Αν υπάρχει θέληση, υπάρχει και τρόπο. Αυτό πιστεύω εγώ. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να επισημάνουμε το πρόβλημα, να πούμε ότι το πρόβλημα είναι η πειρατεία και πρέπει να στραφούμε και στα κράτη-μέλη και στην Κομισιόν που έχουν ζητήσει να υπάρχει ασφάλεια δικαίου κτλ και να δούμε τι προτάσει έχουν να κάνουν. Αν όχι, ε, αν δεν έχουν να μα πούν τίποτα, εντάξει, συμφωνώ. Αλλά αυτή τη στιγμή να πάρουμε αυτή την απόφαση δεν με βρίσκει σύμφωνο γιατί νομίζω ότι επικεντρωνόμαστε σε λάθο πρόβλημα. Ο Νικολό Ρινάλντι τώρα έχει το λόγο. Απ' την άλλη, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Την προηγούμενη εβδομάδα η ομάδα μα την Πέμπτη το απόγευμα στο Στρασβούργο είχε και πάλι μια πολύ ενδελεχή συζήτηση για την Άκτα. Μας ανησυχεί πάρα πολύ η συμφωνία αυτή. Η ανάγκη της ε, καταπολέμησης, της απομίμησης και της ε, παραποίησης. Αλλά θα πρέπει η ομάδα μας να μείνει ενωμένη και γι' αυτό αντιμετωπίζουμε το θέμα με έναν τρόπο βαθμιαίο θα έλεγα, προοδευτικό. Αποφασίσαμε να καταψηφίσουμε την ε, άκτα, δηλαδή ουσιαστικά να απορρίψουμε τη συμφωνία αυτή άρα να στηρίξουμε τη θέση του εισηγητή. Βέβαια στο βαθμό γιατί αυτή ήταν η συμφωνία, γιατί σήμερα είχαμε μία συνέντευξη τύπου με επικεφαλής τον Γκίφερ Χόφστατ παρουσία όλων των σκιωδών της Άλντε στις διάφορες επιτροπές, καθώς και άτομα που κατά το παρελθόν ήταν πάρα πολύ επικοδομητικά και είχαν θετική προσέγγιση προς τη συμφωνία αυτή και ζητούμε με αυτή την ανακοίνωσή μας από την Κομισιόν να αποσύρει τη συμφωνία, αλλιώς θα την καταψηφίσουμε, είναι σαφές αυτό. Υπήρξε μια επιλογή που την προηγούμενη εβδομάδα συζητήσαμε, ε, να μην ζητήσουμε αναδιαπραγμάτευση της άκτα. Αυτό που θα ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι να αναζητήσει νέα εντολή για κλαδικές συμφωνίες, τομιακές συμφωνίες για καταπολέμηση της απομίμης παραποίησης με διαφορετικά μέσα και εργαλεία, τα οποία θεωρούμε ότι θα είναι πιο ενδεδειγμένος τρόπος αντιμετώπισης του προβλήματος από ό,τι με την άκτα. Αν θέλετε μπορώ να επεκταθώ και να σας αναφέρω πιο αναλυτικά τι συζητήσαμε εσωτερικά στην ομάδα μου, πάντως αυτή είναι η θέση στην οποία καταλήξαμε. Και νομίζω ότι είναι γνωστά σε όλες τα επιχειρήματα. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Επόμενος, David Campbell. Είναι εδώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ας ξεκινήσω λέγοντας πρώτα απ' όλα ότι επειδή εγώ γράφω ε, script για ταινίες, έχουν ενδιαφέρον όχι όμως χρηματικό. Εγώ θέλω να προστατευτούν τα δικαιώματα δημιουργού. Δεν θα, θέλω, δεν θα ήθελα ποτέ οι ταινίε εγώ που φτιάχνω το script, ε, ε, να, το σενάριο να πολλούνται πάμφθηνα ε, στο διαδίκτυο από εδώ και από εκεί. Τι γίνεται όμως με την πρόσβαση. Φυσικά και όλοι θέλουμε να υπάρχει η κατάλληλη προστασία από την πειρατεία, αλλά ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες. Ωραία έκφραση είναι αυτή. Και τι συμβαίνει τελικά. Όλοι είμαστε δυσαρεστημένοι με μεγάλο μέρος του κειμένου και το επίπεδο λεπτομέρειας ε, της άκτα. Έχω κάποιες ερωτήσεις. Αν απορριφθεί αυτό το κείμενο, τι γίνεται με την άκτα. Συνεχίζονται διαπραγματεύσεις ή πεθαίνουμε και πεθαίνει και το θάβουμε το πράγμα. Δεύτερο ερώτημα, αν η Ευρωπαϊκή Ένωση απορρίψει την άκτα, αλλά η Αυστραλία ή δεν ξέρω κάποιο προς τη συμφωνία, την υπογράψει. Τι θα έχουμε τότε. Θα έχουμε ένα είδος ε, φυγής ε, όλων των ανθρώπων οι οποίοι ε, θα φύγουν από την Ένωση και θα πάνε στη ΣΥΠΑ ή στην Αυστραλία. Νομίζω θα ήταν καταστροφικό αν κάποιοι κρίνουν ότι ε, δεν μπορούν ε, πλέον να είναι προστατευμένοι εδώ, θα πάνε κάπου αλλού. Αυτά που είπε ο David Martin είναι πολύ σημαντικά, γιατί είναι σημαντικά ζητήματα για τις οικονομίες μας και για, τις, ε, για του Βασιλείου. Χρειάζονται λοιπόν διασφαλίσεις από πολλές εκλογικές περιφέρειες και από την αλληλογραφία που λαμβάνω ακούω συχνά ότι ναι, θέλουμε προστασία και καλύτερη προστασία, αλλά δεν είμαστε πεπισμένοι ότι αυτό θα το πετύχει άκτα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε Τώρα η πράσινη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, θα μιλήσω στα σουηδικά. Στην δική μας πολιτική ομάδα χαιρετίσουμε το γεγονός ότι αποφάσισε ο Ντέιβιτ Μάρτιν να απευθύνει αυτή τη σύσταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευθύς εξ αρχή ήταν ε, σαφές ότι υπήρξαν προβλήματα διαφάνειας σε σχέση με την άκτα. Και εμείς ε, πάντοτε ε, προειδοποίησαμε λέγοντας ότι οι διαπραγματεύσεις πηγαίνουν στην εσφαλμένη κατεύθυνση και δεν ε, παρέχεται ουσιώδης και αποτελεσματική προστασία με τον τρόπο αυτό. Το ζητούμενο ήταν να δούμε τι θα γίνει μελλοντικά όσον αφορά την ελευθερία έκφρασης, τις δημοκρατικές ελευθερίες, αλλά και την αντιμετώπιση των αντίστοιχων αγορών. Οι πράσινοι θα υπερψηφίσουν. Πιστεύουμε ότι είναι καλό που ο εισηγητής προσπάθησε να βρει νέες λύσεις για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ε, ε, ενδεχομένως θα μπορούσαμε να προβάλλουμε κάποιες άλλες λύσεις, διαφορετικές από αυτές που προτείνει ο εισηγητής στο δικό του κείμενο. Αλλά εν γέννη συμφωνούμε μαζί του. Και εμείς κατ' ουσία θεωρούμε επίσης ότι χρειαζόμαστε μια μεταρρύθμιση των εσωτερικών συμφωνιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και όσον αφορά τις συμφωνίες με τους άλλους ε, φορείς, με τους άλλους παράγοντες. Χαιρόμαστε που ο Ντέβιτ Μάρτιν ε, ζητεί την επιβολή κυρώσεων στην περίπτωση παραβιάσεων στις ε, δραστηριότητες στο διαδίκτυο. Θα πρέπει να υποθεί εντελώς ξεκάθαρα το ποια θα πρέπει να είναι η δομή της συμφωνίας, το ποια είναι η δομή της συμφωνίας. Δηλαδή το γεγονό ότι εμεί θέλουμε να προστατευτούν οι πολίτε, ούτω ώστε να μην υπάρχουν ανεπιθύμητε επιπτώσει για να μην ε, οδεύσουν τα πάντα προ μια ασφαλμένη κατεύθυνση. Ε, σε ευχαριστούμε θερμά, Ντέιβιτ, σε ευχαριστούμε θερμά για την εργασία σου. Thank you. Ευχαριστούμε. Και τώρα θα ανοίξει συζήτηση με τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής ή από μέλη άλλων επιτροπών. Υπάρχουν πολλά αιτήματα. Θα θέσω λοιπόν μια, ένα όριο τριών λεπτών για τον κάθε ομιλή. Ο κύριος Λάγκε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Την τελευταία εβδομάδα οι σοσιαλιστές οι και δημοκράτες ε, συζήτησαν την πρόταση του David Μάρτιν και μπορώ να σας πω ότι στηρίζουμε με μεγάλη πλειοψηφία την πρόταση του David Μάρτιν. Δηλαδή πρόκειται να υπερψηφίσουμε την έκθεση κατά της ΑΚΤΑ. Ε, αναλύσαμε επακριβώς την ε, συμφωνία και θα ήθελα συμπληρωματικά προς τα είπε ο κύριος Μάρτιν να αναφερθώ σε δύο σημεία. Όταν μιλούμε για την άκτα συζητούμε για κάποιο συγκεκριμένο αριθμό χώρων και αυτοί που είναι η βασικοί αίτια της πειρατείας δεν συγκαταλέγονται μεταξύ αυτών. Αυτό είναι το σημείο κριτικής. Δηλαδή αυτός ο διαμοιρασμός, ο διαχωρισμός μεταξύ προβάτων και ρηφίων δεν είναι ορθός. Αγαπητοί συνάδελφοι, υπάρχουν και άλλοι που πλήττονται, αλλά δεν μπορούν να πούνε ή όχι στην άκτα. Για παράδειγμα, γενώσιμα φάρμακα τα οποία τα κρατούν στους λιμένες της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρόλο που δεν προορίζονται για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήδη τώρα γίνεται κάτι τέτοιο και δεν θα πρέπει να ενισχύσουμε αυτές τις τάσεις μέσω μιας τέτοιας συμφωνίας, αλλά αντιθέτως θα πρέπει να προσπαθήσουμε σε διεθνές επίπεδο να συνάψουμε λογικές συμφωνίες που να περιλαμβάνουν όλες τις χώρες. Άρα λοιπόν υπό την έννοια αυτή η άκτα δεν θα επιφέρει καμία πρόοδο, αντίθετα θα εδρεώσει ένα εσφαλμένο στάτους κβο ε, και θα επιφέρει, συνεπιφέρει ακόμα περισσότερα προβλήματα. Ποια είναι αυτά τα προβλήματα. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι στιγμής ε, δεν έχουμε μια λογική αντιμετώπιση του προβλήματος πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο. Είναι πραγματικά διεστραμμένο να κάνουμε μια τέτοια συμφωνία και όταν έρθει η Κομισιόν με μία πρόταση για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων στο διαδίκτυο, τότε να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε πώς μπορούμε να το εξασφαλίσουμε. Νομίζω ότι θα πρέπει να βρούμε αποτελεσματικές ε, μορφές προστασίας των ε, δικαιωμάτων αυτών στην Ευρώπη για το διαδίκτυο και στη συνέχεια να περάσουμε στις άλλες χώρες, αυτό που γίνεται παγκοσμίω. Στη Γερμανία υπάρχει μια ολόκληρη βιομηχανία κατά της ε, ε, κακής ε, κατά της εκμετάλλευσης φωτογραφιών, για παράδειγμα στο Facebook. Επιβάλλονται πρόστιμα από αυτούς τους τιμωρούς των παραβιάσεων στο διαδίκτυο. Αλλά δεν είναι δυνατόν να ισχύσει, να αφήσουμε να ισχύει αυτή η κατάσταση. Θα πρέπει να αναλάβουμε εμεί τις ευθύνες μας. Ο κύριος Ζαλεύσκη από το ΕΛΚ έχει το λόγο. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ τον ε, εισηγητή, ο οποίος ε, δείχνει ότι η προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων είναι πολύ σημαντικό θέμα και ταυτόχρονα αποφασίζει να μην στηρίξει την άκτα και να αυτή τη σύσταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, τονίστηκαν διάφορες ε, πτυχές που εγείρουν κάποιες αμφιβολίες και θα πρέπει να γίνουν αντικείμενο μιας νέας διαπραγμάτευσης. Και νομίζω ότι αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή, γιατί η άκτα ε, κατέδειξε ένα πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα από τα προβλήματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Ε, κατέδειξε ότι το μοντέλο αυτοπροστασίας της ε, πνευματικής ιδιοκτησίας, το οποίο κληρονομήσαμε από το 19ο αιώνα και τη Σύμβαση της Βέρνης, δεν ενδείκνυται πλέον για τον 20ο αιώνα, όπου έχουμε το διακδίκτυο και μια ολόκληρη επανάσταση στον χώρο της ανταλλαγής απόψεων και άρα συνεπώς θα πρέπει να προσαρμόσουμε την νομοθεσία μας σε αυτή τη νέα λογική η οποία ε, όπως ε, κατανοώ δεν ε, ελήφθη ευθύς εξ αρχής υπόψη. Δεν επικρίνουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά την ΑΚΤΑ. Το αρχικό project ήταν εντελώς απαράδεκτο και δεν μπορούσε να ευθυγραμμιστεί με τη δική μας νομοθεσία. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπάθησε να ξεφορτωθεί αυτά τα αρνητικά στοιχεία, αλλά δυστυχώς δεν το πέτυχε. Ε, αυτή τη στιγμή η άκτα είναι νεκρή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να την αποσύρει. Δεν έχει απολύτω κανένα νόημα να συνεχίσει τι προσπάθειέ τη να την περάσει. Συμφωνώ με, τη, με τον κύριο Λάγκε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έπρεπε να προετοιμάσει μια νέα πρόταση όσον αφορά την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων, επεκτείνοντα τι λεγόμενε επιτρεπτέ χρήσει, allowed uses. Και στη συνέχεια αυτή η νέα, το νέο μοντέλο θα πρέπει να συμπεριληφθεί στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Και μόνο τότε θα ξεκινήσουμε να διαπραγματευόμεθα ένα καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας για το ίντερνετ. Νομίζω ότι οι προτάσεις της Άλντε να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας ε, μπορεί να γίνει δεκτή, πιστεύω. Και νομίζω ότι το αποτέλεσμα έχει ως εξής. Η άκτα θα πρέπει να αποσυρθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα πρέπει να προετοιμάσουμε ένα νέο μοντέλο copyright, επεκτείνοντας σε επιτροπές χρήση στο διαδίκτυο και μόνο στη συνέχεια θα πρέπει να ξεκινήσουμε διεθνείς διαπραγματεύσεις για να προστατεύσουμε αυτό το νέο μοντέλο των πνευματικών δικαιωμάτων. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Θα τηρήσω τα χρονικά περιθώρια. Καταρχήν ε, πιστεύω ότι το επίπεδο κριτικών κατά των συμπερασμάτων των συντονιστών να καταψηφιστεί η άκτα ε, δεν είναι απολύτως ορθές. Γιατί οι συντονιστές κατέκτησαν σαφές ότι δεν είναι η αρχή της ε, παραποίησης της ε, πνευματικής ιδιοκτησίας η οποία ε, διακυβεύεται στη δική, στην γνωμοδότησή τους. Αλλά είπαν ότι υπάρχει αμοιβαία συμφωνία από όλες τις ομάδες για την βασική αυτή αρχή. Και το βασικό επιχείρημα είναι ότι ο νόμος όσος έχει, η συνθήκη όσο έχει, προσπαθεί καταρχήν να κάνει υπερβολικά πολλά πράγματα ενσωματώνοντας διαφορετικά στοιχεία, ετερογενή στοιχεία και κάνοντας μια αναλογία μεταξύ, ε, φυσικής, ε, μεταξύ υλικής κλοπής και πνευματικής κλοπής, πράγματα που ε, δεν είναι ταυτόσιμα. Δεύτερον, είναι μια παράνομη συνθήκη η οποία προσπαθεί να καταπολεμήσει την παραποίηση και ε, γι' αυτό σε μια ποινική διαδικασία κάποιος θα πρέπει να έχει απολύτως ξεκάθαρες ε, γραμμές. Και αν ε, η ίδια η κλοπή δεν ορίζεται επακριβώς, αλλά αναφέρεται σαν μια εμπορική δραστηριότητα ή σαν μια εμπορική πράξη, τότε στις περιπτώσεις αυτές, με ένα πολύ απλό παράδειγμα, ο Ντέιβιτ δημιούργησε ή γύρε κάποιες αμφιβολίες όσον αφορά την απλούστατη των πράξεων. Ε, για παράδειγμα, ε, καταγγέλλοντας ε, τον συνάδελφο ο οποίος θέτει ένα συγκεκριμένο θέμα σε σχέση με τον συνάδελφο και του το μεταθέτει και καταλήγει σε μια τέτοιου τύπου ποινικοποίηση όπως αυτή που αναφέρει η συνθήκη. Το θέμα είναι ότι θα μπορούσε να είναι μεγάλο επίτευγμα αν αυτή η συγκεκριμένη συνθήκη ε, μπορούσε να περάσει γιατί καλύπτει 50% του παγκόσμιου εμπορίου. Αυτό είναι το βασικό επιχείρημα, αλλά είναι παραπλανητικό αυτό το επιχείρημα γιατί δεν είναι το, το ποσοστό συγγνώμη, του παγκοσμίου εμπορίου που θα πρέπει να εκτιμηθεί, αλλά το ποσοστό της πειρατεία εντός αυτού του εμπορίου. Εάν η πλειοψηφία της πειρατεία γίνεται εκτός αυτού του 50%, στην περίπτωση αυτή και μεταξύ χωρών που παραβιάζουν τον νόμο, τότε ο νόμος είναι ε, ε, λάθος, εσφαλμένος. Άρα λοιπόν δεν είναι σωστό να πούμε ότι καλύτερα να έχουμε κάτι από το να μην έχουμε τίποτα και αυτό το κάτι καλύπτει το 50%. Δεν είναι σωστό αυτό το επιχείρημα. Το επιχείρημα θα πρέπει να είναι, και καταλήγω εδώ, ότι η πειρατεία εντός αυτού του 50% είναι 40%. Ε, συγγνώμη, η πειρατεία είναι, ε, γίνεται μεταξύ των χωρών εκείνων που δεν πρόκειται να υπογράψουν αυτή τη συνθήκη. Simon Κύριος Μπουσούντιλ, τώρα από την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ και από το ΕΛΚΑ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ναι, πράγματι είμαι από την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, άρα υπό αυτό το πρίσμα βλέπω τα πράγματα. Θα ξέρετε ότι η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών προετοιμάζει γνωμοδότηση υπό το άρθρο 36 του κανονισμού που λέει κατά βάση ότι η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών μπορεί να προετοιμάζει μια γνωμοδότηση για να λέξει κατά πόσον ένα έγγραφο, ένα νομοθέτα με μια συνθήκη συνάδει με ε, τα νομοθεσία για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Έχουμε προγραμματίσει και αύριο μια συνάντηση για την ΑΚΤΑ. Όταν εγκριθεί η γνωμοδότησή μα, στη συνέχεια υποχρεωτικά θα επισυναυτεί, θα προσαρτηθεί στην έκθεση τη καθήλυνα αρμόδια επιτροπή, της επιτροπής ΣΥΝΤΑ δηλαδή, στην προκειμένη περίπτωση. Φαίνεται σαφέ, αν και ακόμη δεν έχουμε τα συμπεράσματα τη Επιτροπή ΛΥΜΠΕ, αλλά φαίνεται σαφέ ότι κάποια προβλήματα πράγματι έχουν εντοπιστεί σε σχέση με την άκτα. Νομίζω δηλαδή ότι πια υπάρχει συμφωνία μεταξύ όλων. Ο επόπτης, ο Ευρωπαίος Επόπτης για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων επίσης έχει επισημάνει σοβαρές ε, δυσκολίες με τη συμφωνία. Το ερώτημα είναι το εξή. Από τη στιγμή που έχουμε βρει δυσκολίε στην άκτα, τι κάνουμε. Καταψηφίζουμε άμεσα τη συμφωνία ή προσπαθούμε να την αλλάξουμε, να την τροποποιήσουμε. Και αυτή είναι η επιλογή που έχουμε να κάνουμε. Πολλοί είπαν ότι ε, πρέπει να σκοτώσουμε την άκτα. Άλλη επιλογή είναι να προσπαθήσουμε να τη διορθώσουμε. συνάδελφο ε, Κέλνερ νομίζω ε, είπε πολλά καλά επιχείρηματα υπέρ τη δεύτερη επιλογή και νομίζω ότι είναι σκόπιμο να ακολουθήσουμε αυτή την προσέγγιση. Πρώτα απ' όλα, μπορούμε να αφαιρέσουμε τα τμήματα που δεν μας αρέσουν και να διατηρήσουμε αυτά που μας αρέσουν. Και έτσι αλλάζει η συμφωνία. Γιατί φαντάζομαι οι συνάδελφοι συμφωνούν ότι πρέπει να καταπολεμηθεί η απομίμηση παραποίηση. Αν βέβαια δεν αλλάξουμε, φυσικά μπορούμε να καταψηφίσουμε. Είμαστε έφερα να καταψηφίσουμε τη συμφωνία. Τουλάχιστον να προσπαθήσουμε να τροποποιήσουμε τη συμφωνία με επικοδομητικό τρόπο, διατηρώντας πάντοτε το δικαίωμά μας να την καταψηφίσουμε όποτε το θελήσουμε. Η διαπραγματευτική μας θέση θα ήταν και ισχυρότερη. Διότι αν απορρίψουμε τη συμφωνία θα πρέπει να ξεκινήσουμε από το μηδέν. Τώρα, με τη συμφωνία PNR για τα δεδομένα των επιβατών, ακριβώς το ίδιο πράγμα κάναμε. Ήρθε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με μια συμφωνία που είχε διαπραγματευτεί με τις ΗΠΑ. Τέτοια εποχή πέρυσι. Όταν είχε υποβάλει αυτή την συμφωνία, η ίδια τη νομική υπηρεσία είχε πει ότι παραβιάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα με τη συμφωνία αυτή. Και τι κάναμε εμεί, ζητήσαμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ξαναπάει και να διαπραγματευτεί τη συμφωνία με τι ΕΠΑ, ώστε να πάψουν να παραβιάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θα μπορούσαμε πέρσι να είχαμε την επιλογή να σκοτώσουμε άμεσα τη συμφωνία PNR. Αντίθετα, επιλέξαμε να ζητήσουμε αναδιαπραγμάτευση. Αυτό έγινε και την προηγούμενη εβδομάδα μόλις εγκρίθηκε η συμφωνία PNR και μάλιστα με στριπτική πλειοψηφία από το Κοινοβούλιο. Ολοκληρώνω λοιπόν, έχουμε επιλογή. Είτε καταψηφίζουμε τώρα, είτε τροποποιούμε τη συμφωνία. Νομίζω ότι η πιο λογική λύση είναι να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε τη συμφωνία. Σας ευχαριστώ πολύ. Τώρα έχει το λόγο ο κύριος Κασπάρη από το ΕΛΚΑ με κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να πω ότι συμφωνώ απολύτως με τους προλαλήσαντες, γιατί πιστεύω ότι συζητούμε όλοι, ε, συμφωνούμε όλοι για τις ε, αδυναμίες της άκτα, αλλά θα πρέπει να είμαστε τίμιοι. Γιατί υπάρχει άκτα. Υπάρχει άκτα γιατί η βασική παραγωγή των παραπαϊπιένων ε, προϊόντων στο πλαίσιο του ΠΟΕ ή άλλων θεσμών δεν ήταν διατεθειμένοι να συζητήσουν μαζί μας για αυτό το θέμα. Και εφόσον έτσι έχει η κατάσταση και έτσι είχε στο παρελθόν, γιατί να αλλάξει αύριο. Δεν έχουμε τέτοιες ενδείξεις. Θα χάσουμε 10, 15, 20 άλλα ακόμα χρόνια ε, στον αγώνα πάταξης της ε, πειρατείας. Αλλά θα χάσουμε χρόνο θα χάσουμε χρόνο όσον αφορά τις θέσεις εργασίας, θα χάσουμε χρόνο όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών μας. Γι' αυτό δεν είναι η σωστή απάντηση να στελιτεύσουμε την άκτα, αλλά θα πρέπει να την επιδιορθώσουμε, όπως είπαν οι προηγούμενοι ομιλητές. Γι' αυτό ε, και γι' αυτό ε, πιστεύω θα πρέπει να παραμείνουμε έντιμοι, ειλικρινοί σε αυτό το κοινοβούλιο. Και όπως έγινε με άλλα μεγάλα προγράμματα, για παράδειγμα στο περιβάλλον, στο πρωτόκολλο του Κιώτο, οι βασικοί ρηπαίνοντες δεν, είναι, δεν ε, συμμετέχουν. Η Κίνα, οι Ηνωμένε Πολιτείε κλπ. Όχι, δεν συμμετέχουν. όλα αυτά, εμείς ε, το κάνουμε γιατί θεωρούμε ότι θα πρέπει κάποιος να κάνει την αρχή, να κάνει τα σωστά βήματα. Και το ίδιο ισχύει και για τα φάρμακα. Βεβαίως είναι ένα πρόβλημα όταν ε, φάρμακα τα οποία ε, ε, χρειάζονται κατεπηγόντως τελικά κατακρατώνται. Ε, το πρόβλημα είναι... Θα ξύνει αυτό το πρόβλημα η άκτα. Όχι, γιατί η άκτα δεν αγορίζεται κατά των φαρμάκων, αλλά κατά των παραποιημένων φαρμάκων. Είναι καλύτερα αγαπητοί συνάδελφοι όταν κάποιοι άρρωστοι στην Αφρική παίρνουν κάποια παραπημένα φάρμακα τα οποία δεν έχουν απολύτως καμία δράση αλλά έχουν μια ωραία συσκευασία και προέρχονται από το κύκλο του οργανωμένου εγκλήματος και οι άνθρωποι τα παίρνουν και πεθαίνουν καλό είναι αυτό. Νομίζω ότι θα είναι καλύτερο να κάνουμε κάποιες σκέψεις σε σχέση με το πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε στους ανθρώπους αυτούς τα σωστά φάρμακα και να πατάξουμε το οργανωμένο έγκλημα. Γι' αυτό, κύριοι συνάδελφοι, εγώ πρόκειται ε, θα πρέπει να διατυπώσουμε ξεκάθαρα τις απόψεις μας, θα πρέπει να δώσουμε και το χρόνο στην Επιτροπή να κάνει τις δικές της σκέψεις. Δεν είναι δυνατόν να τσαλακώσουμε, να καταπατήσουμε τα πάντα, να τσαλαπατήσουμε τα πάντα και να αρχίσουμε από μηδενική βάση. Δεν είναι δυνατόν αυτό να αποκληθεί υπεύθυνη πολιτική. Finally Δεν χρειάζεται να επαναλάβω τα όσα είπα. Είναι η πρώτη φορά που συζητάμε το θέμα αυτό εκτός από το workshop, το εργαστήριο. Ξέρετε ότι εγώ είμαι υποστηρικτής της άκτα, δεν χρειάζεται να το επαναλάβω. Τα επιχειρήματα είναι γνωστά. Γι' αυτό θέλω να θέσω δύο ερωτήσεις. Μία προς το ίδιο το κοινοβούλιο, σε εμά. Νομικός είναι δυνατόν, πολιτικός είναι επιτρεπτόν να ψηφίσουμε μια διεθνή συμφωνία που είναι υπό εξέταση από το ΔΕΚ. Ξέρετε ότι η Κομισιόν έχει στείλει αυτή την ε, συμφωνία στο ΔΕΚ που και του ζητά να εκρευνήσει αν είναι μόρφη προς τις συνθήκες και το χάρη των θεμελιωδών δικαιωμάτων ή όχι. Όποια και αν είναι η μελλοντική απόφαση του δικαστηρίου, Δεν μπορούμε να ψηφίσουμε κάτι που ενδέχεται το δικαστήριο να το θεωρήσει ε, παράνομο ή μη σύμμορφο προς συνθήκες. Πάντως χρειάζεται να διευκρινιστεί. Δεύτερο ερώτημα είναι το εξής. Είναι σαφές ότι ότι η συμφωνία άκτα θα απορριφθεί από το Κοινοβούλιο και αν γίνει αυτό το ερώτημά μου είναι προς την Κομισιόν. Έχει η Κομισιόν κάποια ιδέα για το πώς ε, θα συμπεριφερθούν τα υπόλοιπα συμβαλόμενα μέρη, η ΕΠΑ και οι υπόλοιποι θα συνεχίσουν και θα μας αφήσουν πίσω ή είναι έτοιμοι να διαπραγματευτούν εκ νέου μία συμφωνία. Δεν είναι διμερή συμφωνία, είναι πολυμερής. Και αυτή η ερώτηση είναι κατά την απόψη μου πολύ σημαντική. Μπορώ να φανταστώ ποια θα είναι η αντίδραση των υπολείπων συμβαλωμένων μερών. Θα, θα προχωρήσουν χωρίς εμάς, αλλά ίσως η Κομισιόνα να έχει κάποια άλλη ερμηνεία για τη... πώς θα κινηθούν οι εταίροι μας. Η πρώτη ερώτηση ξέρετε από εμά. Η δεύτερη θα ήθελα να ακούσω την απάντηση της Κομισιόν. Δίνω λοιπόν το λόγο στην Κομισιόν, τον κύριο Μασάντο. To the Council representative. Uh, και έπειτα στον εκπρόσωπο του Συμβουλίου. Τον εκπρόσωπο της Δανικής Προεδρίας. Κύριε Μασάντο, έχετε το λόγο. Δεν μπορώ να σας δώσω και άπειρο χρόνο. Έχουμε 25 λεπτά στη θέση μας. Πρέπει και ο να πει την τελευταία λέξη, να συνάγει τα συμπεράσματά του. Κύριε Γιγέρμα Σάντο, λοιπόν, όχι πάνω από 7 λεπτά. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είμαι ευτυχής που έχω την ευκαιρία να ανταλλάξω απόψεις μαζί σας για αυτή τη σημαντική συνθήκη που έχει δώσει δηλαδή για πολλές ε, πολεμικές και διαφορετικές ε, και υπάρχουν πολλές διαφορετικές απόψεις. ήθελα να ξεκινήσω αναγνωρίζοντας αυτό που αναγνωρίζει και η έκθεση και ο εισηγητής ότι το άκτα ή η συμφωνία άκτα ασχολείται με ένα πραγματικό και ε, υπαρκτό πρόβλημα που είναι η παραβίαση των ευρωπαϊκών πνευματικών δικαιωμάτων. Πρόκειται για τε μεγάλες ε, κλίμακες δραστηριότητε, για μεγάλη ζημιά για την οικονομία μας που θέτει σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια ε, των Ευρωπαίων πολιτών. Όπως γνωρίζετε στην Ευρώπη έχουμε ένα συνολικό σύστημα για την προστασία και την επιβολή της πνευματικής ιδιοκτησίας. Έχουμε περιγράψει τα δικαιώματα που μπορούν να προστατευτούν και τα μέσα για την επιβολή αυτών των δικαιωμάτων. Έχουμε εφαρμόσει αυτό το σύστημα στα κράτη-μέλη μαζί με τις εθνικές αρχές. Όταν διαπραγματευθήκαμε το σύστημα για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων στην Ένωση, επιλέξαμε να διατηρήσουμε το δικαίωμα των πολιτών στην ελεύθερη έκφραση, την προστασία των στοιχείων και την πρόσβαση στις πληροφορίες, καθώς και το δικαίωμα των ε, προμηθευτών ε, υπηρεσιών ίντερνετ και άλλων διαμεσολαβητών να μπορούν να προσφέρουν αυτά τα αγαθά. Αυτοί οι δύο στόχοι είναι συμβατοί και αλληλοϊποστηριζόμενοι αμοιβαίω. Αυτό επιτύχαμε με το ΙΝΑΚΤΑ. Αυτό που προσπαθεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση με αυτή τη συμφωνία είναι να επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής αυτού του τμήματος αυτού του συστήματος των ευρωπαϊκών νομοτικών δικαιωμάτων και της προστασίας τους πέρα από τα σύνορά μας. Εκείνο το τμήμα που θέλουμε να προστατεύσουμε είναι οι διαδικασίες για την επιβολή και όχι τα δικαιώματα αυτά καθ' αυτά. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό να τονιστεί. Η άκτα δεν λογοκρίνει το ίντερνετ. Δεν επιβάλλει υποχρεωτικό έλεγχο η παρακολούθηση των, ε, της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του κόσμου. Δεν μπλοκάρει οποιαδήποτε δραστηριότητα ανταλλαγής πληροφοριών, αλλά ούτε και επιβάλλει ε, περιορισμούς στο εμπόριο των, ε, γεν... των... Ε, των γενώσιμων φαρμάκων είναι φτιαγμένη, κομμένη και ραμμένη με βάση το ευρωπαϊκό σύστημα ώστε να μπορούμε να κάνουμε και υπάρχει δυνατότητα τροποποίησης της ισχύουσας νομοθεσίας. Αυτό σημαίνει πως η άκτα δεν θα έχει οποιασδήποτε μη ε, προβλεπόμενες ε, συνέπειες. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό γιατί δεν ε, θα θίγει την βασική ευρωπαϊκή νομοθεσία. Οι περισσότερες ανησυχίες που ακούμε περί της άκτα φαίνεται να βασίζονται στην, πίστη, στην άποψη ότι οι δικαιούχοι δικαιωμάτων μπορούν άμεσα να επιτεθούν κατά της άκτα κατά μεμονωμένων καταναλωτών. Αυτό δεν είναι δυνατόν. Είναι αδύνατον. Αυτό που ισχύει και θα συνεχίσει να ισχύει για τους Ευρωπαίους πολίτες δεν είναι η άκτα, αλλά ο κοινοτικός νόμος. Η άκτα δεν θα είναι άμεσα εφαρμόσιμη στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι μόνοι κανόνες που θα ισχύσουν είναι αυτοί που ήδη υπάρχουν μέσα στο κοινοτικό κεκτημένο και θα εξακολουθήσουν να ισχύουν με η άνευ άκτα. Οποιαδήποτε αλλαγή για αυτούς τους κανόνες θα πρέπει να περάσει από το Κοινοβούλιο και οι Ευρωπαίοι καταναλωτές πάντοτε θα προστατεύονται από τον Ευρωπαϊκό νόμο. Και εδώ ε, θίγω ένα τα ερωτήματα που τέθησαν που ήταν το ότι θα πρέπει να περιμένουμε την Κομισιόν για τις νέες προτάσεις για την προστασία των δικαιωμάτων. Εδώ δεν έχουμε θέμα γιατί το ένα δεν αποκλεί το άλλο γιατί το άκτα δεν ασχολείται με τα δικαιώματα αυτά καθ' αυτά όπως σας είπα. Ασχολείται με την επιβολή αυτών και την προστασία αυτών. Αυτό δεν εμποδίζει λοιπόν η Ένωση και το Κοινοβούλιο να εξετάσουν μελλοντικέ προτάσεις και να αλλάξουν και το κοινοτικό κεκτημένο. Η συμφωνία άκτα αφορά μόνο την επιβολή και οι ουσιαστικές διατάξεις ε, βρίσκονται αλλού. Επίσης έχουμε υπόψη ότι δεν προβλέπεται μηχανισμός ρύθμισης διαφορών. Η ερμηνεία των κανόνων της ΑΚΤΑ θα ελέγχονται από την ίδια την Ένωση. Το επιχείρημα δηλαδή ότι η εμπορική κλίμακα στι διατάξει ΣΑΚΤΑ είναι αόριστο και ότι υπάρχει κίνδυνο η δικιά μα ερμηνεία τη Ένωση να είναι σε κίνδυνο γιατί άλλοι θα το ερμηνεύσουν διαφορετικά, δεν έχει νόημα γιατί δεν υπάρχει κανόνα. Δεν υπάρχει, προβλέπεται μάλλον μηχανισμός ρύθμισης, δεν υπάρχει δηλαδή ε, διαιτητικός μηχανισμός στη μέση. Αυτό είναι το παράδειγμα που μόλις έδωσα και που είναι ένας, μια από τις επικρίσεις που ακούσαμε ε, σε σχέση με το, την εμπορική κλίμακα, ότι δηλαδή αυτός ο όρος είναι πολύ ανακριβής. Αλλά πέρα από τον κίνδυνο που σας περιέγραψα ήδη, ότι δηλαδή δεν μπορεί κανείς να μας επιβάλλει οτιδήποτε όσον αφορά τα δικαιώματα ε, ε, δεν υπάρχει γιατί αυτή η κλίμακα ήδη ισχύει εδώ και πολλά χρόνια και ισχύει σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία. Ε, έχει εφαρμοστεί από τα δικαστήριά μας σε χιλιάδες περιπτώσεις και θα συνεχίσει να ισχύει σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία άσχετα από την άκτα. Η υποχρέωση ε, ποινικοποίησης της πειρατείας των πνευματικών δικαιωμάτων ήδη ισχύει επίσης και ήδη εφαρμόζεται από τις περισσότερες χώρες παγκοσμίω. Τη μεγάλη πλειοψηφία των κρατών μελών του ΠΟΕ και τα λοιπά. Η άκτα περιλαμβάνει ε, μέτρα ποινική επιβολή μόνο για πολύ σοβαρέ παραφιάσει που έγιναν ηθελημένα και σε εμπορική κλίμακα. Αυτό το κριτήριο της εμπορική κλίμακας είναι πολύ σημαντικό και ξέρω πως δεν έχουμε χρόνο, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να αυτά τα κριτήρια να ερμηνεύονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο ξεκάθαρα. Ξέρω ότι τελειώνει ο χρόνος. Θέλω σύντομα να αναφερθώ στα, ερωτήσει ερωτήσεις που θέσατε. Τι θα γίνει αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απορρίψει τη συμφωνία. Τότε η Ένωση δεν θα ε, συνυπογράψει συμφωνία. Πρέπει να ε, εγκριθεί από το Κοινοβούλιο και από το Συμβούλιο. Γιατί δεν το κάνουμε μέσω του ΠΟΕ. Και αυτή είναι η καλή πρόταση. Το προσπαθήσαμε και το προσπαθεί η Ένωση εδώ και πολλά χρόνια. Αλλά εκεί δεν έχουμε βρει υποστηρικτέ. Και έπειτα Υπάρχει και το εξή ε, επιχείρημα ότι δεν έχουμε το σωστό στόχο μέσω τη άκτα γιατί οι περισσότεροι μεγαλύτερο όγκο πειρατεία, δηλαδή οι βασικέ χώρε που παράγουν πειρατικά αγαθά, δεν είναι μέλη τη άκτα. Το 50% μάλλον είναι εκτό. Εντάξει, μπορεί να. Ναι, όντω. Η Κίνα δεν είναι μέσα και πολλοί που παράγουν παραποιημένα ή πλαστά αγαθά δεν το υπογράφουν. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε πως αυτές οι χώρες πουλάνε αυτά τα πλαστά προϊόντα στι ανεπτυγμένε αγορέ, Δηλαδή, Ένωση, ΙΠΑ, Ιαπωνία. Δηλαδή τις χώρες που είναι συνυπογράφοντα μέλη τη ΑΚΤΑ. Αφού παράγουν και πάνε να πει ότι πουλούν και που πουλούν στις αγορές μας. Έπειτα, ο ισχυρισμό ότι προκαλεί απειλή, ότι αποτελεί απειλή, για τα θεμελιώδη δικαιώματα. Νομίζω πως αυτός ο ισχυρισμός είναι πολύ σοβαρός και πρέπει να αποφασιστεί από το αρμόδιο όργανο, δηλαδή το ΔΕΚ. Και γι' αυτό και στραφήκαμε σε αυτό. Και ο καλύτερος τρόπος είναι να περιμένουμε την απόφαση του Συμβουλίου, του δικαστηρίου με συγχωρείτε, πριν να προβούμε σε λήψη απόφασης. Και ακούσουμε και το Συμβούλιο, να κλέψουμε λίγα λεπτά, γιατί τα κάλυψε η Κομισιόν. Ποιος θα μιλήσει από πλευρά του Συμβουλίου. που πρέπει να επικυρωθεί όχι μόνο από την Ένωση αλλά και από τα κράτη-μέλη, γιατί είναι οι υπηρεσίες εδώ. Τα κράτη-μέλη που είναι μέλη του Συμβουλίου. Τι γίνεται λοιπόν, το Συμβούλιο μπορεί να μας πει ποια είναι η κατάσταση όσον αφορά την επικύρωση σε εθνικό επίπεδο. Well, um, ε, κύριε Πρόεδρε, πρώτα απ' όλα, Πρόεδρε, αγαπητοί βουλευτές, η Προεδρία χαίρεται που της τη δυνατότητα να συμμετέχει στις εργασίες της Επιτροπής σας ε, για την Συμφωνία Άκτα για να σας παρουσιάσουμε τις απόψεις μας σχετικά. Η Προεδρία αντιλαμβάνεται πλήρως την ευαισθησία του θέματος και τον σημαντικών ανησυχιών που έχουν εκφραστεί και από την κοινή γνώμη αλλά και από βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων που συνεδρίασε στις 16 ε, Μαρτίου ενημερώθηκε για την πρόθεση της Κομισιόν να παραπέμψει την άκτα στο δικαστήριο που θα πρέπει να αποφαθεί για το κατά πόσον ε, είναι συμβατό η συμφωνία με την συνθήκη, συγκεκριμένα για τις θεμελιώδεις ελευθερίες, ελευθερία έκφρασης, πληροφόρησης, προστασία δεδομένων, δικαίωμα ιδιοκτησίας, συγκεκριμένα σε περίπτωση πνευματικής ιδιοκτησίας. Στις 4 Απριλίου η Κομισιόν επισήμως αποφάσισε να υποβάλει νομίμως ε, την άκτα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο λόγω των ε, ευρυτάτων ανησυχιών και προβλημάτων που είχαν προκύψει. Το Συμβούλιο έχει ρετήσει την απόφαση της Κομισιόν να παραπέμψει το θέμα της άκτα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο είναι σε μια μοναδική θέση για να αποφανθεί κατά πόσο η άκτα συνάδει με τις συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Συμβούλιο προσβλέπει με ανυπομονησία στην ετοιμιγορία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου αφού το δικαστήριο είχε, θα έχει αρκετό χρόνο για να εξετάσει εντελεχώς την υπόθεση και να συνεισφέρει μετά στην διαδικασία. Για το ερώτημά σας, να σας ενημερώσω ότι η υπογραφή της ΑΚΤΑ συμφωνήθηκε ομόφωνα από τα μέλη του Συμβουλίου στις 16 Δεκεμβρίου του 2011. Έχει οργανωθεί στο Τόκιο για τον Ιανουάριο του 2012 υπογραφή της συμφωνίας. Δεδομένης της ανάγκης ε, να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες εσωτερικές διαδικασίες ώστε οι εκπρόσωποι να εξουσιοδοτηθούν μόνο 22 κράτη-μέλη ήταν στην ε, υπογραφή. Τα υπόλοιπα πέντε κράτη μας είπαν ότι θα προχωρήσουν στην υπογραφή όταν ολοκληρωθούν οι εθνικές τους, οι εσωτερικές τους διαδικασίες και η Προεδρία βέβαια είναι σε επαφή με τα λίγο κράτη-μέλη. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Thank you very much. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο εισηγητής, έχετε το λόγο για τα τελικά συμπεράσματα μετά από αυτήν την πολύ καλή συζήτηση. Ναι, ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρέπει να πω ότι δεν είναι η πρώτη φορά που έχω απορρίσει, αλλά όχι από τα άλλα θεσμικά όργανα, από την Επιτροπή μας. Πραγματικά διερωτώ με αν οι συνάδελφοι ε, κατάλαβαν την αρχική μου πρόταση, που ήταν αυτή, να πάμε στο 10 και ότι κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου εγώ θα έκανα μια διάμεση έκθεση που θα εξέταζε κάθε τμήμα για το τι σημαίνουν τα μέτρα, να ζητώσω από την Επιτροπή τι είδου οδηγίε θα στείλουμε στου προμηθευτέ των υπηρεσιών να του ζητήσουμε τον ορισμό τη εμπορική κλίμακα και το απορρίπτασατε. Και ωστόσο, τέσσερι συνάδελφοι που είχαν καταψηφίσει εκείνη την πρόταση έρχονται σήμερα και μου λένε ότι πρέπει να δούμε πιο λεπτομερό στην άκτα και να πάρουμε λίγο περισσότερο καιρό για να φτάσουμε σε συμπεράσματα. Αυτό ήταν το αρχικό μου επιχείρημα. Το κάναμε και εγώ ε, έφαγα τα μούτρα μου τότε. Ε, τώρα πρέπει όμως να λάβουμε μια απόφαση. Και αν λάβουμε απόφαση, και αυτή η ερώτηση είναι τμήμα της απάντησης, και αν η απόφαση είναι όχι στο, στην άκτα. Η απόφαση λέει ότι αν έξι υπογράψουν την άκτα θα συνεχίσει, θα προχωρήσει μάλλον, το 42 της συμφωνίας επιτρέπει την νέα διαπραγμάτευση. Ε, μπορούν δηλαδή να επανέλθουν τα κράτη-μέλη και να προτείνουν και τροποποίηση στη συμφωνία. Ίσως λοιπόν και δεν ε, σας συστήνω αυτή την πορεία, αλλά μπορεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να πει όχι και είμαστε σαφείς για το γιατί λέμε όχι. Η Κομισιόν μπορεί να θέλει να επανέλθει στους υπόλοιπους, στα συμβαλόμενα μέλη και να ξεκινήσουν μια τροποποιητική διαδικασία. Μπορεί δηλαδή να υπάρξει ένα σενάριο όπως με τα στοιχεία των ε, επιβατών αεροπορικών εταιριών και το σημαντικό είναι ότι όπως έχουν τα πράγματα, εμείς θα πρέπει να καταψηφίσουμε τη συμφωνία. Ωραία. Για τέλος της συνεδρίασής μας για σήμερα. Ε, υποβολή τροπολογιών και προθεσμία για την υποβολή. Θα έχουμε την 10η Ιουνίου, μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Δεν έχουμε κάτι άλλο για απόψε. Αύριο θα τα πούμε και θα συνεχίσουμε στις 9 το πρωί. Ευχαριστώ πολύ.